Εσύ για να μην καθυστερήσουμε ανώφελα. Θα σας παρακαλέσω να ξεκινήσουμε λοιπόν. Καλωσορίζω τους πάντες και ενημερώνω ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στην εμερήσια διάταξη πλην μίας. Ότι δηλαδή ο κύριος Ράσφαν Κούργεναρου θα έρθει για την κυρία Ελένα Ουντρέα, την Υπουργό. Θα έρθει ο Ήφη Υπουργός από τη Ρουμανία. Ιδάλω αλλαγή δεν υπάρχει στην ημερήσια διάταξη από πλευρά μου. Επίση σα ενημερώνω ότι ω ήθιστε μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μα. και αν δεν υπάρχουν σχόλια στην ημερήσια διάταξη θα περάσω στο σημείο 2, έγκριση των πρακτικών τη συνεδριάσεω μα 21 και 22 Μαρτίου. Και πάλι ως ήθιστα έχετε τα πρακτικά στη διαθεσή σας, έχουν διανεμηθεί τα πρακτικά. Και άρα στο τέλος συνεδρίας, αν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις, θα θεωρηθεί ότι εγκρίθηκαν. Παρακαλώ. Κυρία Μανέσκου. Ακούστε. Ναι, καλημέρα πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να μπορούμε, ε, ακριβώ να μπορέσουμε να δεχτούμε μια συζήτηση για μια ανταλλαγή απόψεων με τον ε, Υπουργό Μουργιάνου ε, αν θα μπορούσαμε να το δεχτούμε και αν ακριβώς Προσκαλέσαμε την κυρία Ούντρα γιατί ο συνάδελφος Λάμπερτ ε, που δεν είναι στην αίθουσα σήμερα εδώ θα ήθελε να προχωρήσουμε σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων με την Υπουργό και όχι με κάποιον άλλο. Εντάξει, θα μπορούσαμε να περιμένουμε και τους συναδέλφους μας, τους συντονιστές, για να τους ρωτήσουμε αν θέλουμε να έχουμε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ θα ήθελα να σας πω ξεκινώντας ότι έχω την ίδια άποψη όπως από τους ελεύθερους την συντονίστρια. Θα ήθελα όμως κυρία Πρόεδρε να προσθέσω κάτι και αγαπητοί συνάδελφοι. Αποφάσισε η Επιτροπή μας να αναβάλει για την εκθεσία αυτή την ψηφοφορία μέχρι να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια συζήτηση με την ε, Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης γιατί υπάρχουν πολλές και σοβαρές, ε, πολλά και σοβαρά θέματα και οι συζητήσεις ε, στη Ρουμανία που συζήτηση που είχαμε με την Υπουργό Εξωτερικών και με ορισμένους υπουργούς όλοι μας περιμέναμε τελικά μια απάντηση η οποία δεν μας ήρθε και ακόμα κυρία Πρόεδρε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η δική μας η Επιτροπή έδειξε κάθε καλή διάθεση ότι θέλαμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά με τις αρχές της Ρουμανίας και ότι θα θέλαμε να τις υποστηρίξουμε τις αρχές της Ρουμανίας ακριβώς για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και την Παρασκευή μας πέρασε μερικά μέλη από τη δική μας επιτροπή πήγαν στο Βουκουρέστι και συμμετείχαν σε μια συνάντηση με την πρόεδρο κ. Ωγνερ και σχετικά με την περιφερειακή μεταρρύθμιση και δυνατότητα απορρόφησης κονδυλίων όπως επίσης και την περιφερειακή ανάπτυξη στη Ρουμανία. Δυστυχώς δεν συμμετείχε τότε η Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης στη συνάντηση αυτή. Βλέπουμε ότι αυτό γίνεται κάτι που επαναλαμβάνεται γιατί ούτε σήμερα δεν συμμετέχει εδώ στη συζήτηση. Γι' αυτό συμφωνώ με την πρόταση κ. Μανέσκου. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να δεξάγουμε μια συζήτηση σχετικά με την κατάσταση όχι μόνο για τα επιχειρησιακά προγράμματα, όπως επίσης και για τα γενικά προβλήματα απορρόφησης των κονδυλίων από τη χώρα αυτή που δυστυχώς ε, από την 1η Μαρτίου είναι στην τελευταία θέση, στη χειρότερη θέση όσον αφορά την απορρόφηση κονδυλίων. Ε, από τη στιγμή που ζητάμε από την υπεύθυνη υπουργό να έρθει εδώ και για, να, για λόγους σεβασμού ακριβώς προς την Επιτροπή μας πρέπει να σέβεται την Επιτροπή μας. Ε, θέλουμε να ενημερωθούμε σχετικά. Και εντάξει, εδώ και 15 χρόνια ε, την γνωρίζω. Δεν πρόκειται για μια αντίθεση απέναντι στην κυρία Μουργιάνου, Αλλά νομίζω ότι η κυρία Υπουργό η ίδια θα πρέπει να παραστεί εδώ και να δείξει την καλή της διάθεση και το σεβασμό της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εδώ, εντάξει, το Εθνικό Κοινοβούλιο... Ε, Υπάρχει ένα μπλοκάρισμα όσον αφορά τις ψηφοφορίε. αλλά όχι εδώ όμω, στη δικιά μα επιτροπή δεν μπορούμε να παίξουμε το ίδιο παιχνίδι και να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Πρόεδρε, ευχαριστώ και στο συγγνώμη που καθυστέρησα λίγο να έρθω στη συνεδρία. Θεωρώ όμω ότι είναι πράγματι πολύ δύσκολο να δεχθούμε το ότι δεν έρχεται η ίδια Υπουργέ να μα ενημερώσει, δεδομένου ότι είναι εδώ στι Βρυξέλλες. Δεν έχω καμία κατανόηση για τη συμπεριφορά αυτή. Εμείς είμαστε εδώ νομοθετικό όργανο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετοιμάζουμε την επόμενη περίοδο. Και θέλουμε να δούμε πώς προχώρησε η Ρουμανία, όπως και τα άλλα κράτη βέβαια, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όντως ξέρουμε ότι η Ρουμανία προξενεί κάποιε ανησυχίες ως προς το ε, ρυθμό απορρόφησης και την ε, εφαρμογή των προγραμμάτων των κονδυλίων δηλαδή στην ε, Ρουμανία, στο εσωτερικό τη. Καλό λοιπόν θα ήταν να έρθει η ίδια η Υπουργός να μας μιλήσει. Εάν αυτό δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ακόμη σήμερα, από ό,τι φαίνεται δεν είναι δυνατόν, καλό θα ήταν να ενημερώσουμε στο Βουκουρέστι ότι περιμένουμε την Υπουργό ενώπιον μας για να λάβει θέση. Και θέλουμε και εξηγήσει γιατί αγνοεί την Επιτροπή μας. Το βρίσκω παράδεκτο αυτό. Ευχαριστώ, Λόχανεν και μετά Φαν Ρόιν, Ή Τούμπαλιν. Λαμπέρ Φαν Νίστελ Ο κύριος Φαν Ναι, εγώ έλαβα τις πληροφορίες τις σχετικές ε, χθες το απόγευμα, 5 η ώρα. Κοιτάξτε, είναι θέμα προοπτικής. Πρώτα απ' όλα, ως επικεφαλής αντιπροσωπείας έχουμε την έκθεσή μας και νομίζω ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε την έκθεση αυτή και να την ολοκληρώσουμε. Παράλληλα, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλή ευκαιρία και για την εξέταση του περιεχομένου, θα ήταν καλό να είχαμε εδώ την Υπουργό, την κυρία Ουντρέα. Εγώ προτείνω να κάνουμε κανονικά τη δουλειά μας, να συνεχίσουμε τη δουλειά μας εξετάζοντας την έκθεση και αν υπάρχει δυνατότητα, αλλά βέβαια αυτό είναι ένα ζήτημα δούνε και λαβίν, γιατί δεν μπορεί κανείς να διατάξει σε κανέναν υπουργό να έρθει ε, σε μια επιτροπή όταν εμείς θέλουμε να έρθει. Αυτό είναι ένα ζήτημα το, οποίο ενδεχομένω θα έπρεπε να υποβάλει η πρόεδρο τη Επιτροπή μα. Όντω. Τουλάχιστον όμω εμεί από τη δική μα πλευρά μπορούμε να συνεχίσουμε με την, εξέ, με την εξέταση της ε, έκθεσή μας παρουσία του ε, εκπροσώπου της Ρουμανίας, ο κύριος Λούχαν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω το σχόλιο του κυρίου Βανίστελ Ρόι. Δεν πιστεύω τώρα εδώ ότι θα πρέπει να μπούμε σε συζητήσεις ποιος θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση σε αυτή τη σημερινή συζήτηση που θα πρέπει να είναι συζήτηση επικοδομητική σχετικά ακριβώς με την έκθεση της Επιτροπής μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δούμε τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες και να δούμε πώς έχει πραγματικά η κατάσταση για την δυνατότητα απορρόφησης κονδυλίων από τη Ρουμανία. Νομίζω ότι αυτό προχωράει καλά, όπως ε, το θεωρώ τουλάχιστον εγώ. Μερικά σχόλια για το τι έγινε τώρα τελευταία, τι εμφανίστηκε στον τύπο της Ρουμανίας. Ορισμένες ενέργειες ε, των συναδέλφων μας από τους φιλελεύθερους για να αποπροσανατολίσουν και μάλιστα το είχαν σαν σκοπό αυτό την κοινή γνώμη τη ρουμανική για να επιτεθούν στην κυβέρνηση της δεξιάς από έχουμε, έχουν συνασπισμό εκεί. Και εδώ σχετικά με τις δραστηριότητες μας ε, δεν θα πρέπει να επικεντρώνουμε την προσοχή μας στο τι συμβαίνει έτσι πολιτικά. Ούτε και λαϊκιστικά να το αντιμετωπίζουμε αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με μια συζήτηση ουσίας και ε, συμφωνώ με την πρόταση του κ. να αναβάλουμε ε, μάλλον ναι, δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ με την πρόταση του κυρίου Στενάρου ε, για την αναβολή αυτή τη συζήτηση επειδή δεν παρίσταται η Υπουργό Περιφερειακή Ανάπτυξη. Ο Ναι, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η ιδιαιτερότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να προσπαθεί να εξεύρει συμβιβασμού και νομίζω. εντάξει, το σημερινό παράδειγμα είναι και ένα ερώτημα που τίθεται για τις επόμενες ε, συνεδριάσεις μας. Ε, μπορούμε να ζητήσουμε να μας ε, αποστείλει μια κυβέρνηση μόνο έναν υπουργό ή κάποιον γενικό από την κυβέρνηση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε γενικότερα για το μέλλον. Μέχρι τώρα, κατά παράδοση, ζητούσαμε κάποιον από, τον από το Υπουργείο και αποφασιζόταν ε, κατά πόσο θα έρθει ο ίδιος ο Υπουργός ή κάποιος άλλος. Καταλαβαίνω βέβαια το ότι ο συμβιβασμός ε, είναι μια απογοήτευση που ανέφερε και η κυρία, κυρία Ρόιλ επειδή ήταν εδώ η Υπουργός, είναι εδώ Υπουργός και δεν μπορεί να ε, παραστεί σήμερα και επομένως έστειλε κάποιον άλλον στη θέση της. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε στο μέλλον. Ίσως θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι όντως μας δυσαρεστεί αυτό, Νομίζω όμως ότι για τις μελλοντικέ μας δραστηριότητες αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να αφήνουμε την απόφαση στην κυβέρνηση σε σχέση με το ποιο θα την εκπροσωπήσει. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλα σχόλια? Αν όχι. Πρώτα κάποιες διευκρινήσεις. Καταρχώς, καταρχάς ναι, πράγματι μπορούμε να καλέσουμε κάποιον από τις ε, μπορούμε να, να καλέσουμε και οι εθνικές αρχές θα αποφασίσουν ποιος είναι ο κατάλληλος για να παραστεί στην συνεδρίασή μας. Εμείς ζητήσαμε βέβαια να έρθει ε, η υπουργό, γιατί αυτή την απόφαση είχαμε λάβει ως ε, Επιτροπή και εγώ έλαβα απέστειλα ότι έλαβα μια επιστολή από την κυρία Ουντρέα ότι ε, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων ζήτησε από τον κύριο Μουργεάνου να την αντικαταστήσει. Αυτό σας το λέω διευκρινιστικά. Δεύτερο ζήτημα. Η έγκριση της έκθεσης ε, της επίσκεψης στη Ρουμανία συνδέθηκε με την συζήτηση που θέλαμε να κάνουμε με την Υπουργό σήμερα και υπάρχει μια πρόταση να μην το αναβάλουμε, αλλά να το συζητήσουμε σήμερα ε, με τον εκπρόσωπο της Ρουμανίας και η άλλη επιλογή βέβαια είναι να αναβάλουμε ε, εντελώς τη συζήτηση, να μην το συζητήσουμε καθόλου. Η πρότασή μου είναι να γίνει ανταλλαγή απόψεων σήμερα σε σχέση με την έκθεσή σας ε, για την επίσκεψη αντιπροσωπείας, παρουσία του κυρίου Μουργιάνου και θα ήθελα να πω ότι θα έρθω σε επαφή με την κυρία Ουντρέα με την Υπουργό για να δω κατά πόσο υπάρχει μια ημερομηνία ε, στην οποία μπορεί να παραστεί στο μέλλον ε, για να έχει αυτή την ανταλλαγή απόψε μαζί μας. Αν θέλετε, μπορούμε να φτάσουμε και ήδη στην ψηφοφορία, αν δεν συμφωνείτε. Ο κύριος Βουστινάρου. Κυρία Πρόεδρε, κοιτάξτε. Εντάξει. Αλλά ένα πράγμα νομίζω πρέπει να το διευκρινίσουμε. Θα μπορούσατε να μας πείτε, κάποιος θα μπορούσε να μας πει στο δωμάτιο, αν η Υπουργό είναι σήμερα στι, στην, ε, στις Βρυξέλλες ή όχι, γιατί αν είναι στις Βρυξέλλες η κυρία Ουντρέα και παρά το γεγονός ότι είναι στις Βρυξέλλες δεν θα παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειών, εγώ το βρίσκω πραγματικά τόσο απαράδεκτο. Εγώ είμαι υπέρ του να συζητήσουμε αυτή την έκθεση για τη Ρουμανία, γιατί είναι σαφέστατα τα συμπεράσματα, αλλά μπορούμε εμείς να αποδεχθούμε ως Επιτροπή η αξιοπιστία μας ε, να αμφισβητείται κατά αυτόν τον τρόπο. Πρόεδρος, κοιτάξτε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι στις Βρυξέλλες η κυρία Υπουργό. Ε, αν θέλει κανείς να πάρει το λόγο και να μας διευκρινίσει το ζήτημα αυτό, ευχαριστώ. So, we don't know. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν. Uh, so there is a proposal. Ο κύριος Μποστινάρου να ρωτήσουμε το γραφείο του Επιτρόπου Χάν για να ξέρουμε κατά πόσα υπάρχει συνεδρίαση σήμερα. Κοιτάξε, Βίκτορ, κοίταξε, Βίκτορ, εγώ λέω να το διευκρινίσουμε αυτό πιο μετά. Έχουμε τώρα προβλέψει στην ημερήσια διάταξή μα χρόνο για τη συζήτηση του θέματο αυτού και πρέπει να αποφασίσουμε κατά πόσο θα κάνουμε την ανταλλαγή απόψεων αυτή τη στιγμή και μετά ε, θα δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα. Λοιπόν, να γίνει μια μικρή παρουσίαση ε, για την έκθεση αυτή και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Ήταν πάρα πολύ ευγενική η επιστολή της κυρίας ε, Ουντρέα και συνδέει την απουσία της με ε, παράγοντες. Λοιπόν, έχουμε ένα ακόμη θέμα στην ημερήσια διάταξη πριν την ανταλλαγή απόψεων για τη Ρουμανία. Ο Λάσλο είναι εδώ να περάσουμε στο 4 της ημερησία διάταξης. Εντολή για τον τριμερή διάλογο. Κύριε Λούχαν, μόνο απλώς να διευκρινίσω κάτι. Εχθές, μία ώρα πριν πω στο αεροπλάνο, μύρισα με την κυρία Υπουργό. Δεν είναι στις Βρυξέλλες σήμερα. Σας το λέω αυτό με βεβαιότητα. Θα ήθελα να ρωτήσω την ε, κυρία Κρόελ να μας πει από πού έχει τις πληροφορίες αυτές ότι είναι εδώ στις Βρυξέλλες. Δεν είναι στις Βρυξέλλες η κυρία Ουντρέα. Της μιλούσα μία ώρα πριν μπω στο αεροπλάνο. Εχθές, πρόεδρος. Ωραία. Υποθέτουμε λοιπόν ότι δεν είναι στις Βρυξέλλες η υπουργό. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Περνάμε στον Λάσλο Σούριαν. Πολύ σύντομα, αν μπορείς Λάσλο να μας κάνει την παρουσίαση. Θυμάσαι ότι είχαμε κάνει μια μεγάλη συζήτηση για το θέμα αυτό την περασμένη φορά. Υπάρχει τίποτε άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις. Έχεις το λόγο. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Να και εγώ είμαι στις Βρυξέλλες τώρα. Ας συνεχίσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό τουλάχιστον. Πολύ σύντομα λοιπόν. Έχουμε ένα κείμενο το οποίο ε, συνοψίζει, ομαδοποιεί σε πέντε σημεία τις προτάσεις μας και προτείνω αυτό να αποσταλεί στην Επιτροπή των προϋπολογισμών, φυσικά με ενσωματωμένες και όποιες πιθανές τροπολογίες. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι, σε αυτό το στάδιο προετοιμασίας του προϋπολογισμού, ότι υποστηρίζουμε την πολιτική συνοχής και όλα τα ε, χρηματοδοτικά μέσα που προβλέπονται για αυτήν και θέλουμε σαφείς δεσμεύσεις για, τα μελλοντικά, για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές. Όπως είπα, δεν έχω ακριβή αριθμητικά στοιχεία σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, αλλά πιστεύω ότι τα πέντε σημεία μας αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες, τα μελήματα τα σχετικά με την, ε, με την πολιτική συνοχής. Και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να το δουν όσοι ασχολούνται με την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Ζητούμε να εφαρμόσετε σε ένα πλαίσιο επταετίας το πρόγραμμα για την πολιτική συνοχής. Έχουμε πληρωμές που βλέπονται υψηλές το 2012 και το 2013, δηλαδή φτάνουμε στην περίοδο εχμής της εφαρμογής αυτής της επταετίας, της τρέχουσας και έτσι πρέπει να στραφούμε και προς την στρατηγική για το 2020 και τη χρηματοδότηση της τελευταία ανάλυση. Οι στόχοι δεν απέχουν πολύ μεταξύ πολιτικής συνοχής και στρατηγικής του 2020. Ε, θα ήθελα ωστόσο να υπογραμμίσω ιδιαίτερα μέσα στο κείμενο ότι δεν είναι και ταυτόσιμοι οι στόχοι. διότι μπορεί να υπάρχει αναφορά στο ποια περιφέρεια Φερρυπίν θα λάβει δυνατότητα υποστήριξη για την ανάπτυξη των θέσεων εργασία, αλλά νομίζω ότι από πλευρά μα εμεί θέλουμε να υποστηρίξουμε την ανάγκη για περισσότερη υποστήριξη των περιφερειών ώστε να φτάσουν στο επίπεδο των πιο προηγμένων. Δεν μπορούμε λοιπόν να εξομοιώσουμε πολιτική συνοχή με στρατηγική τη Λισαβόνα ή ακόμη και να υπαγάγουμε την πολιτική συνοχή να την εντάξουμε δηλαδή εξ ολοκλήρου μέσα στη στρατηγική της Λισαβόνας. Πρέπει όμως να βρούμε την, τα σημεία της επαφής και τα σημεία που μπορούν να λειτουργήσουν συνεργατικά οι δύο αυτές πολιτικές. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι έχουμε κοινή ευθύνη έναντι του Ευρωπαίου φορολογουμένου ως προς την διάθεση των απαραίτητων, των αναγκαίων κονδυλίων με ένα χρονοδιάγραμμα προσεκτικά προετοιμασμένο και πιστεύω ότι κάθε φορά που βλέπουμε υπουργό εδώ στην Επιτροπή μας θα πρέπει να, τους να τον ενθαρρύνουμε ε, να προχωρήσει περισσότερο σε αυτή την εφαρμογή. Η πιο καθυστερημένες περιφέρειες δηλαδή, οι πόλεις, θα πρέπει να έχουν και αυτές την ευκαιρία να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Σε αυτό θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Θα ήθελα να πω ότι για τη δική μου την περιοχή, στην Ουγγαρία, έχουν τριπλασιαστεί οι προκαταβολές τελευταία περίοδο, πράγμα το οποίο δείχνει ότι όταν υπάρχει επαρκής επιμέλεια και φροντίδα ε, προσεκτική προετοιμασία και εκτέλεση από πλευρά του κράτους μέλους βελτιώνονται κατά πολύ οι επιδόσεις. Θέλουμε λοιπόν και την απλούστευση στην εφαρμογή, όπω ζητάει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χωρί να θέλω λοιπόν να σα καθυστερήσω περισσότερο, θα ήθελα να υπογραμμίσω ορισμένα σημεία για το χρονοδιάγραμμα και ε, συγκεκριμένα για τις 14 Απριλίου, αυτή την εβδομάδα ακόμη, την Πέμπτη, έχουμε προθεσμία για την κατάθεση ανθρωπολογίων για το πολύ σύντομο αυτό κείμενο. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, λέει ο κ. Σούζαν και έχουμε συνεδρίαση το Μάιο 24 και 25 αν δεν απατώμε οπότε και θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε τότε φαντάζομαι την έκθεση θα πρότεινα για την προσεχή εβδομάδα 20 Απριλίου που πρόκειται να υπάρξει ε, ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκεί δηλαδή θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για το 2012 και θα πρότεινα ω συντονιστή τη Επιτροπή μα για τα θέματα του προπολογισμού να συμμετάσχω εγώ στη συνεδρίαση αυτή, όπου θα δημοσιευθεί η ανακοίνωση από τον Επίτροπο και ίσω να προτείνω ω εισηγητή σχετικέ τροπολογίε στο κείμενό μου. Φυσικά δεν μπορώ τώρα να προεξοφλήσω εάν αυτοί, αυτές οι τροπολογίες που πιθανώς ε, ε, καταθέσω θα είναι υπέρ της ανακοινώσεως επιτροπής εάν αντιθέτως θα σας προτείνω να ε, προβούμε σε διορθώσεις του κειμένου της ανακοίνωσης. Πάντως, διορθώσεις θα είναι δυνατές φαντάζομαι, όπως πάντοτε υπήρχε η δυνατότητα. Θα είμαι σε επαφή πάντα με τους συντονιστές και ό,τι προτάσεις, ό,τι τροπολογίες θα είμαι στη θέση για να τις ενσωματώσω στο κείμενό μου, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Λάσλο και τώρα να ακούσουμε τους σκιώδεις συγγητάς, παρακαλώ. Όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Έχουμε καθυστερήσει πολύ. Και μην λησμονούμε ότι έχουμε συζητήσει ήδη. Πριν από τρει εβδομάδε συζητήσαμε το θέμα αυτό. Ο κύριο Βόν, λοιπόν, πρώτο. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ ιδιαίτερα στον εισηγητή για την έκθεση. Είναι σύντομη, είναι εύστοχη και συμπεριλαμβάνει και αρκετές καλές προτάσεις. Εν γέννη συμφωνώ με τον εισηγητή ότι η πολιτική συνοχής είναι απαραίτητη για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά σε μια χρονική περίοδο που χρειαζόμαστε ε, και θέσει εργασίας και ανάπτυξη. Για την υπαριθμόν ένα παράγραφο θα ήθελα να επισημάνω τα προγράμματα για το 2007-2013 πλέον φτάνουν στην ε, ταχύτητα κρουαζιέρας όπως λέμε και κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε και τη μέγιστη απορρόφηση των κονδυλίων ή τουλάχιστον κατανομή των κονδυλίων. Έχουμε φτάσει τουλάχιστον δική μου την περιφέρεια στο 80%. Και νομίζω ότι στο 2 προσπαθεί ο εισηγητής να επισημάνει ότι είναι αποδεκτή η στόχη της στρατηγικής του 2020 αλλά δεν μπορεί να είναι η μόνη μας στόχη. Σε αυτό επίσης συμφωνώ. Έχουμε διαφορετικ... Έχουν διαφορετικές προτεραιότητες ε, η μεν και η δε και γι' αυτό θα έπρεπε ναι, να πούμε ότι υπάρχουν κοινά σημεία, σημεία επαφής αλλά οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές. Για να καταλήξω λοιπόν, θα περάσω τώρα στην παράγραφη παριθμών όπου πιστεύω συμφωνούμε όλοι πως χρειάζονται επαρκείς και κατάλληλοι πόροι για την επιτεύξη του στόχου της συνοχής, της πολιτικής της συνοχής, πολύ σωστά, αλλά μια και φτάνουμε στην περίοδο αυτή της ε, ταχύτητας κρουαζιέρας, ίσως θα έπρεπε να αναζητήσουμε περισσότερου πόρου, να εξασφαλίσουμε περισσότερου πόρου για την πολιτική συνοχή στον προπολογισμό για το 2012. Και αυτό θα μπορούσαμε να το ενσωματώσουμε στην, στην πέμπτη παράγραφο. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Θέλει κανεί να λάβει το λόγο. Καλώ, ο κύριο Αλφονσί. Κυρία Πρόεδρε, γρήγορα, γρήγορα εγκρίνομαι τις ε, βάσεις αυτής της έκθεσης ε, και για το ενδιαφέρον της Επιτροπής Προλογισμού ότι πρέπει κάθε χρόνο να βλέπουμε πιστώσεις πληρωμών υψηλότερε γιατί φτάνουμε ακριβώς σε αυτή τη φάση που πραγματοποιούνται αυτά τα εφαρμόζονται αυτά τα προγράμματα και αν ε, το αναβάλουμε αυτό τότε θα αναχαιτιστεί όλη η κατάσταση αυτό λοιπόν και θα ήθελα επίσης εδώ μιλάμε για τις διαδικασίες που να είναι πιο απλές και ένα ερώτημα γιατί γίνεται με τα σχέδια πιλότους μήπως ε, θεωρεί ότι κάτι θα πρέπει να προβλεφθεί ώστε να ληφθούν αυτά τα σχέδια υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Πατρίς Αγαπητοί συνάδελφοι, μέχρι το 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει 200, ε, τη 272η περιφέρεια και στη Μαγιότ ε, θα είναι υπερπόντια κτήση ακριβώς Γαλλία σύμφωνα με το 355 άρθρο της συνθήκης που προβλέπει κάτι τέτοιο μετά από ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου και αντίθετα με τις τρίτες χώρες δεν υπάρχει κανένα μέσο προένταξης. Θα πρέπει να έχουμε το υψηλότερο επίπεδο απορρόφησης κονδυλίων στην περιφέρεια αυτή από το ξεκίνημα της επόμενης περίοδου προγραμματισμού. Θεωρώ λοιπόν απαραίτητο από του χρόνου και μετά να υπάρξει ένα εργαλείο που θα μπορέσει να προετοιμάσει από τεχνικής κυρίως πλευράς την εφαρμογή της προσεχούς πολιτικής συνοχής. Η Επιτροπή Περφεκής Ανάπτυξης που είναι η άμεσα εμπλεγμένη και υπεύθυνη σε αυτή την ε, σε αυτό που θα συμβεί ακριβώς. Θα πρέπει να το κάνει αυτό στο Κοινοβούλιο στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης περί προϋπολογισμού. Ευχαριστώ για την προσοχή που μου αφιερώσετε. Ευχαριστώ. Κανείς άλλος. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Λάσλο αν θέλει να σχολιάσει ή όχι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω την εντύπωση ότι για παράδειγμα αυτό που είπε ο σοσιαλιστής και ο εισηγητής ε, είναι ακριβώς και ο στόχος του κειμένου. Μπορεί να, μπορούμε να αλλάξουμε λίγο τη διατύπωση, αλλά εγώ αυτό που ήθελα να εκφράσω είναι ακριβώς αυτό, ακριβώς, αυτό ακριβώς που είπε ο, ο συνάδελφος και που ανέφεραν και άλλοι ομιλητές. Τώρα όσον αφορά νεότερες περιφέρειες ε, οι οποίες θα ενταχθούν ε, με τα γενέστερα, Όταν θα φτάσουμε σε εκείνη τη χρονική στιγμή θα δούμε τι θα κάνουμε. Αφόσον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ημερήσια διάταξη αυτό το θέμα, δεν υπάρχει λόγος να κινητοποιήσουμε και ε, μεγάλα ποσά. Δεν ανέφερα επίση στην παρουσίασή μου ότι τα πιλωτικά προγράμματα είναι εξαιρετική σημασίας και πρέπει να μάθουμε και από το παρελθόν. Πέρσι, αν ε, είναι σωστά τα έγγραφά μου, Είχαμε 20 προτάσεις, 6 ήταν επιτυχείς και είναι στο σημερινό προϋπολογισμό, έχουν ενταχθεί στο σημερινό προϋπολογισμό. Αν ε, κάποιος είχε, ήταν ε, νικητής ε, την περασμένη χρονιά, θα ήθελα να μας πει τι έγινε από απόψεως προπαρασκευαστικής και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά εμείς, εγώ ως εισηγητής, έχω σκοπό να συνεχίσουμε με, το, με την προσπάθεια αυτή. Θα είναι η συνήθις προτεραιότητά μου και για το μέλλον. Τα νέα πιλωτικά προγράμματα πρέπει να είναι έτοιμα κανονικά μέχρι το Μάιο έτοιμα για να τα υποβάλουμε στην κυρία Παλτζάνη και να γίνει και ένας προκαταρκτικός έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζετε ότι αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Αν λοιπόν οι προτάσεις σας είναι έτοιμες, παρακαλώ να τις υποβάλλετε το συντομότερο δυνατό. Και αν είχατε την καλοσύνη να με ενημερώσετε και εμένα για τα σχέδιά σας, ε, με πολύ χαρά θα σας ακούσω. Θα αναμένω λοιπόν τις τροπολογίες και ακούγοντας οδη συζητητής είμαι σίγουρος ότι θα τύχει ιδιαίτερη αποτοχή ε, το κείμενο αυτό στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο. Ε, μπορούμε να προσκαλέσουμε και κάποιον από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μα δώσει συνολικά για τα πιλωτικά προγράμματα κάποιε πληροφορίε. Ε, να συζητήσουμε, Λάσλο, ποια θα ήταν η καλύτερη χρονική στιγμή να το κάνουμε αυτό. Το μόνο που έχουμε να αποφασίσουμε σήμερα είναι την προθεσμία για τις τροπολογίες. 15 Απριλίου προτείνω εγώ, 12 η ώρα το μεσημέρι. 15 Απριλίου. Μία ακόμη μέρα δηλαδή, μία παραπάνω μέρα σε σχέση με αυτή που έχεις προτείνει εσύ. Προτείνω λοιπόν να ζητήσουμε από τον ε, κύριο Μουργιάνου να μας, πει, ε, να κάνει μια παρουσίαση και μετά ε, ο επικεφαλής αντιπροσωπείας της επίσκεψης στη Ρουμανία να μας κάνει μια μικρή παρουσίαση και εκείνος και να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων μετά. We start with um, State Secretary uh, Razvan uh, Αρχίζουμε λοιπόν με τον κύριο Μουργιάνου. Oh, Ευχαριστώ, χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που είμαι εδώ, γιατί είστε μία από τις σημαντικότερες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεύτερον, θα ήθελα να σας πω ότι εκπροσωπώ το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Τουρισμού και μπορώ να συζητήσω μόνο ε, το ε, περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα που είναι περίπου 90% ε, της συνολικής χρηματοδότησης για τη Ρουμανία από το 2007 έως το 2013. Θα ήθελα λοιπόν ε, να είμαι πάρα πολύ σαφής ε, για ε, το τι ακριβώς μπορώ να σας συζητήσω μόνο, να σας, να σας να συζητήσουμε σήμερα, όχι για το σύνολο της χώρας μου, αλλά μόνο για το ROP, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Για να δούμε το πρόγραμμα αυτό εφαρμογής είναι το περιφερειακό πρόγραμμα που είναι το 19% αυτής της περίοδου στην Ρουμανία η εξέλιξη αυτού του επιχειρησιακού προγράμματος που σέβεται το σχεδιασμό του 2007 όταν αυτό το πρόγραμμα εγκρίθηκε όσον αφορά τις συμφωνίες και τις πληρωμές. Οι πληρωμές που έγιναν στο περιφερειακό πρόγραμμα ακριβώ οι συνολικές είναι το, Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με συγχρηματοδότηση από την προϋπολογισμό της χώρας μέχρι την 1η Απριλίου του 2011. 3.551.000 λέει και το 20% του προϋπολογισμού είναι του ΦΕΝΤΕΡ για το 2007 στο 2013. Το Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης στις δηλώσεις της Επιτρο... κυβέρνησης είναι 330 εκατομμύριο και είναι 9,1% του προπολογισμού. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως έλεγα λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τις πληρωμές είναι 248 εκατομμύρια ευρώ και είναι το 6,7% του προϋπολογισμού 2007-2013 καταβάλλεται από την Επιτροπή. Μέχρι το τέλος του 2011 η αρμόδια αρχή για την περιφερειακή ανάπτυξη ακριβώς είχε σαν στόχους τους εξής. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και οι δηλώσεις για τις ε, πληρωμές 735 ε, εκατομμύρια ευρώ που είναι το 19,8% των προγραμμάτων. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε, Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν οι διερμηνείς να παρακολουθήσουν αυτή την ταχύτητα δεν μπορούν να παρακολουθήσουν. Διαβάζει νούμερο ο Υπουργό ε, με μια ταχύτητα αδιανόητη. Εάν έχετε του καταλόγου αυτού, ε, του πίνακε, δώστε του στου διερμηνεί να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το νούμερο που εκφωνείτε. Ναι, με συγχωρείτε. Βέβαια, όλα αυτά τα δεδομένα είναι δημόσια. Και θα σας τα στείλω και στην Επιτροπή σας και σε όλους σας τα δεδομένα αυτά, γραπτός, πολύ σύντομα. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερική ανάπτυξη ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν 648 εκατομμύρια ευρώ που είναι το 18,2% του προπολογισμού για το πρόγραμμα αυτό για τα σχέδια που είχαμε στα πλαίσια αυτά. Το σύνολο του επιχειρικού σου προγράμματος του για το 2007-2013 102,74 εκατομμύρια λέει 4 δισεκατομμύρια ευρώ στα πλαίσια αυτά και το σύνολο των συμφωνιών που έκλεισαν μέχρι τώρα 1231 σχέδια, προγράμματα ε, και η συνολική αξία, η συνολική τιμή είναι 14,1 εκατομμύρια 3 δισεκατομμύρια ευρώ, λέει ο Από το ξεκίνημα του προγράμματος ε, αυτά που συμφωνήθηκαν 9,1 εκατομμύρια λέει συγγνώμη αλλά της αριθμός όχι υπουργός 2 εκατομμύρια ευρώ που είναι το 60% περίπου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης από το 2007 μέχρι το 2013. Θα ήθελα να ανοίξω μια σύντομη παρένθεση εδώ. Τη χρονιά αυτή θα τελειώσουμε με το κλείσιμο συμφωνιών όσον αφορά το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα. Όπως έχει ο σημερινός ρυθμός, ε, θα να σας πούμε ότι ενδεχόμενα το Σεπτέμβριο θα ολοκληρωθεί η, θα περάσει η περίοδος για το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα έχουμε 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την όλη διαχείριση. Τα σχέδια όμως ξεπερνούν τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως σας το είπα, είναι σχεδόν τριπλάσια η αξία τους. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης για αυτά τα σχέδια που παρουσιάστηκαν από την αρχή μέχρι σήμερα είναι περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ, 211 περίπου εκατομμύρια στα πλαίσια αυτά. Δυστυχώς, δυστυχώς εμείς ε, μπορούμε να έχουμε μόνο το 150% όχι παραπάνω για την έγκριση αλλά όταν περνάμε από το 150% και πάνω δεν μπορούμε να υποβάλουμε περαιτέρω προγράμματα και ούτε αυτά μπορούν να αξιολογηθούν για να πραγματοποιηθούν ή όχι. Όταν εργαζόμαστε με, με την τοπική διοίκηση το κριτήριο αυτό τι δημιούργησε οι τοπικές αρχές ε, θα ήθελαν να υποβάλουν περισσότερα προγράμματα αλλά το είχαμε τέσσερις μόνο συμφωνίες για 42 δισεκατομμύρια ευρώ παλιότερα τώρα το Μάρτιο του 2011 έχουμε 3 δισεκατομμύρια ευρώ τα κονδύλια που ανέφερα προηγουμένως σχετικά με τα σχέδια αυτά, με τα προγράμματα αυτά. Υπάρχει μια ιδιαίτερη αύξηση και εντάξει μπορώ να μιλάω για αυτά τα στοιχεία προέρχομαι από την τοπική διοίκηση και νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ στην περιφερειακή ανάπτυξη της Ρουμανίας το σχέδιο για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε καλύτερα τα κονδύλια από το Διαθωτικό ατομία και το Ταμείο Συνοχής. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απίφθινε στον Ρουμάνο Πρόεδρο και Πρωθυπουργό μια επιστολή για την μειωμένη δυνατότητα απορρόφησης κονδυλίων της Ρουμανίας και είχε προτείνει δύο κύρια μέσα για την αύξηση της δυνατότητας απορρόφησης. Πρώτα απ' όλα ορισμένα έκτακτα μέτρα, ένα παρόμοιο σχέδιο για περισσότερη απορρόφηση και επίσης ο ορισμός ενός εθνικού συντονιστού υψηλού επίπεδου για αυτά τα ειδικά μέτρα και για την εφαρμογή τους. Και είχαμε πει στην Περιφερειακή Επιτροπή ότι χρειαζόταν ένα σχέδιο με μια εκτίμηση συγκεκριμένη των διαφόρων προβλημάτων και με συγκεκριμένα μέτρα και με ιδιαίτερες ευθύνες από συγκεκριμένα άτομα και επίσης επιμείναμε ε, ότι θα πρέπει να έχουμε διαρθωτικά μέτρα να μπορέσουμε να ελέγξουμε την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Και η αρχή ξεκίνησε τη, να εργάζεται το Φεβρουάριο του 2011 με ένα σχέδιο εθνικών μέτρων ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες ενέργειες για την απορρόφηση αυτών των κονδυλίων στη Ρουμανία. Πρώτη εναλλακτική δυνατότητα η οποία συζητήθηκε μαζί σας στην ετήσια συνάντηση της 3 Φεβρουαρίου φέτος. Υπήρξε και μία αναθεώρηση μετά από παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 3 Μαρτίου πήγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις 15 Μαρτίου ε, προχωρήσαμε και σε σχόλια από ρωμανικής πλευράς για όλα αυτά που συζητήσατε εδώ. Εδώ το τέλος Απριλίου φέτος θα ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία για τις ε, ενέργειες αυτές, για την εφαρμογή του προγράμματος. Ε, η κυβέρνηση της 17 Μαρτίου ε, είπε ότι η σχετική αρχή εργαζόταν κάτω από την ε, έλεγχο τον άμεσο του Πρωθυπουργού και το πρόγραμμα ακριβώς ε, παρουσίαζε το βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα ήθελε να εφαρμόσει η Ρουμανία σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο γενικός στόχος είναι να λυθούν προβλήματα όπως και ανεπάρκειες που έχουν να κάνουν με το σχέδιο εφαρμογής ε, ακριβώς αυτών των προγραμμάτων και για να μειωθούν αυτές οι ανεπάρκειες όσο γίνεται περισσότερο και έχουμε 7 κύριες κατευθύνσεις ε, δραστηριοτήτων και ξεκινώντας από τη σημερινή ανάλυση είδαμε ποια είναι τα κύρια μέσα για να μειωθούν ή για να παλιφθούν τα εμπόδια σχετικά με την απορρόφηση αυτή που παρεμποδίζουν την απορρόφηση. Η διαχείριση του σχεδίου για τα όσα γίνονται από τις ε, αρμόδιες αρχές και οι δημοσιονομικές πτυχές σχετικά με τα επιχειρησιακά προγράμματα και σχέδια Επίση, οι συμφωνίε από κρατική πλευρά και διάφορα άλλα στοιχεία, οι διάφορε δραστηριότητε, οι ελεγκτικέ που είναι και αυτέ άλλο μέσο, η επάρκεια της όλη διαδικασία και όλα αυτά που επηρεάζουν τα πράγματα σχετικά με την εφαρμογή, με την ρύθμιση όλου αυτού του σχεδίου και επίσης διοικητική δυνατότητα ε, απορρόφησης ε, σύμφωνα με προγράμματα που να είναι επιχειρησιακά πραγματικά και δυνατότητα έχουν, έχουν άμεση ευθύνη και οι ωφελούμενοι από τα μέτρα αυτά. Θα πρέπει να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις σύντομα για να πετύχουμε το στόχο ο οποίος έχει τεθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Αναφοράς 2007-2013. Χρειάζεται τουλάχιστον 1% να υπάρξει δυνατότητα απορρόφησης από πλευράς Ρουμανίας. Για το 2011 έστω και ορισμένα μέτρα θα έχουν ε, εν μέρη μόνο εφαρμογή, θα πρέπει να πετύχουμε αυτόν τον φιλόδοξο στόχο, ώστε την τριετία 2012-2015 να μειωθούν όσο γίνεται περισσότερο τα εμπόδια που αναφέρθηκαν. Στο τέλος του 2011 η δυνατότητα απορρόφησης για τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα είναι υψηλότερος, θα αυξηθεί δυνατότητα απορρόφησης κατά 20-25% σε σχέση με το άμεσο παρελθόν. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Λάμπερτ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας έδωσε ο Υφυπουργός. Είχα την ευκαιρία προσωπικώς πρέπει να πω να επισκεφθώ τη Ρουμανία και να συναντήσω αρμοδίους σε διάφορα επίπεδα πολιτικά, να συζητήσω και σε περιφερειακό αλλά και σε τοπικό επίπεδο με εκπροσώπους τοπικών και περιφερειακών αρχών σε διάφορες περιοχές της χώρας Ουσιαστικά κάθε γωνιά της Ρουμανίας επισκέφθηκα. είδα και δομές ε, κοινωνικές, ε, κοινωνικής υποστήριξης Φερρυπίν προς τους Ρώμα για μια μόνιμη εγκατάσταση ε, δομές για την ε, περιβαλλοντικών συνθήκων. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη αυτή που πραγματοποιήσαμε στη Ρουμανία και συστήσαμε πολλά θέματα από αυτά που ανέφερε και τώρα ο κύριος Υπουργό Φερρυπίν, το χαμηλό επίπεδο απορρόφησης. Προσπαθήσαμε λοιπόν ε, στην επίσκεψη αυτή να εντοπίσουμε τους λόγους της χαμηλής απορρόφησης. Είπαμε ότι ίσως να φταίει η χρηματοδότηση ε, ίσως εκεί να υπάρχει δυσκολία, δηλαδή ίσως κάποιες διοικητικές δομές να παρουσιάσουν βραδύτητα ως προς την λειτουργία τους. Μας πιστεύω κάναμε ένα κατάλογο, μια απογραφή των προβλημάτων και πάντως μπορέσαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση στη χώρα. Πάντως διαπιστώνουμε σαφή βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι πολύ καλύτερη αντιμετώπιση των δυσκολιών στη Ρουμανία από ό,τι στο παρελθόν. Βέβαια, στα μέτρα αυτά, τις προτεραιότητες που ανέφερε και ο κύριος Υφυπουργός στα 7 σημεία, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να τοποθετηθεί κανείς κατά τρόπο ε, απόλυτο, δηλαδή να πούμε τα προγράμματα αυτά ή εκείνα επέτρεψαν σε αυτόν ή εκείνο τον βαθμό την τάδε πρόοδο. Αυτό είναι δύσκολο ακόμα να το πούμε, αλλά πάντως μπορούμε να συνεχίσουμε γιατί ήδη μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει γίνει σοβαρή δουλειά με στόχο την βελτίωση της διαχείρισης και ίσως θα μπορούσα καταλήγοντας να σας πω ε, μια ιδέα για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και μπρος στην Επιτροπή. Ε, λίγο χρόνο έχω, το ξέρω, αλλά πολύ σύντομα. Ε, μια και τα ανέφερε ο κύριος Υπουργός. Φέρει πίν, συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών. είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στα προγράμματα αυτά, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει κατακαιρματισμός των τοπικών και περιφερειακών δομών στη Ρουμανία. Πράγμα το οποίο είναι λυπηρό, διότι αν συγκριθεί μάλιστα με την κατάσταση της Πολωνίας, σημειώνεται στο θέμα αυτό συγκεκριμένα καθυστέρηση στην διαχείριση σε διοικητικό επίπεδο. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει απουσία συνοχής ή συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων διοικητικών δομών. Το διαπιστώνουμε αυτό από την επίσκεψή μας στη Ρουμανία. Επίσης, ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει η κατάσταση των Ρωμά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσής τους. Έτσι λοιπόν, εάν δούμε τι είδους χρήματα ε, ορίστηκαν ε, για την κατασκευή μόνιμων κατοικιών για τους Ρωμά, βλέπουμε πάλι ότι υπάρχει πρόβλημα προς την απορρόφηση. Ξέρουμε ότι ο νομοθέτης και διάφορες περιφέρειες, αρκετές περιφέρειες, κυρίως η τιμή Φερρυπίν, θέλουν να προχωρήσουν, θέλουν να βελτιώσουν σοβαρά την κατάσταση για τους Ρωμά με βελτίωση και προγραμμάτων εκπαιδευτικών και με προσφορά προγραμμάτων για την απασχόληση, αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις σοβαρές. Εν πάση περιπτώσει, η υποδοχή που μας επεφύλαξαν ήταν πολύ φιλική. Είδαμε σημαντική πρόοδο, αλλά θα θέλαμε μια πιο λεπτομερή παρουσίαση του προγράμματος ε, υλοποίησης. Γιατί βλέπουμε ότι λέτε κύριε Υφυπουργέ ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρχών της Ρουμανίας στις προτεραιότητες αυτές, τις δράσεις προτεραιότητας, αλλά θα θέλαμε η Επιτροπή να είναι σε θέση να συνομιλήσει με τους διαφόρους εκπροσώπους στα διάφορα επίπεδα από τη Ρουμανία, έτσι ώστε αυτή η αρχή να μετατρέπεται σε συγκεκριμένες δράσεις και να μετατραπεί ιδιαίτερα για την περίοδο 2015 μέχρι 2020 σε συγκεκριμένες δράσεις και κυρίως στον τομέα της συνοχής. Όλα αυτά για να δούμε συγκεκριμένα μέτρα. Θέλουμε να βελτιωθεί λοιπόν η απορρόφηση της χρηματοδότησης ε, για τις ε, δημόσιες αγορές θα πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ρουμανία, αφορά ολόκληρο τον πληθυσμό της ε, ε, όλη τη χώρα. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι ναι μεν τώρα μπορεί να μην έχουμε χρόνο 10 παρα 5 η ώρα να συζητήσουμε διεξοδικά όλα αυτά τα θέματα αλλά πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνήσουν η Επιτροπή με τη Ρουμανία και τις αρχές της Ρουμανίας και αυτό όλο να μετατραπεί σε πράξεις αυτό περιμένουμε να δούμε. Άλλωστε και η έκθεση ξεκάθαρα διατυπώνει την ευχή αυτή για συγκεκριμένες δράσεις, για προτεραιότητες και πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη θέσή μας, έστω και αν δεν είναι τα πιο ευχάριστα στοιχεία αυτά που βλέπουμε, τα ιδεώδη, αλλά θα μπορούσαμε όπως και να έχει να τα χρησιμοποιήσουμε ως μια βάση για να προχωρήσουμε. Αυτό ελπίζω τουλάχιστον, αυτό επιθυμώ. Σας ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Η κυρία Κρέλ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δυστυχώ. Εγώ δεν μπόρεσα να έρθω στην αποστολή αυτή στη Ρουμανία, στο ταξίδι αυτό, αλλά βέβαια τα τελευταία χρόνια έχω επισκεφθεί πολλές φορές τη χώρα και θα ήθελα να πω ότι φυσικά έχουμε εξαίρετα παραδείγματα αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων στη Ρουμανία, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ωστόσο, μεγάλη απόκληση διαπιστώνεται μεταξύ ορισμένων πολύ καλών σχεδίων και προτάσεων και των τεράστιων αναγκών σε υποδομές, σε επενδύσεις υποδομών και σε μάλιστα σε κάθε τομέα υποδομών, είτε πρόκειται για τις μεταφορές, είτε πρόκειται για τις ε, τηλεπικοινωνίες, τη δημόσια υγεία, την εκπαίδευση, τα πάντα. Ανησυχώ πολύ λοιπόν τα κονδύλια τα οποία είναι διαθέσιμα και για τα οποία ο Ευρωπαίος Φορολογούμενος περιμένει μια ορθολογική αξιοποίηση, φοβούμαι ότι ενδέχεται να μην αξιοποιηθούν όπως πρέπει και να χρειαστεί να επιστρέψουν στα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Γι' αυτό λοιπόν επισημαίνω δύο προβλήματα. Μπορεί αυτό να οφείλεται στο ότι υπάρχουν ε, μεν κάποιοι στη διοίκηση, ε, στις διοικητικές δομές οι οποίοι έχουν μια καλύτερη κατάρτιση αλλά εντωμεταξύ αποχωρούν από το δημόσια διοίκηση για να βρουν καλύτερες θέσεις εργασίας και είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν καλύτερα να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια ενδεχομένως και θα ήθελα επίση να πω στον ε, Λάμπερτ ότι έχει δίκιο γιατί εάν εμεί τώρα ρωτάμε τι γίνεται από το 2014 εν ώψη των νέων δημοσιονομικών προοπτικών και τι είδου χρήματα θα έχουμε στα στιγμή για την πολιτική τη συνοχή ή με τι άλλο και όχι μόνο για τη Ρουμανία αλλά για όλα τα κράτη θα πρέπει να είμαστε θέση να αποδείξουμε ότι εδώ έχουμε εξασφαλίσει όχι μόνο από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διατύπωση ωραίων ιδεών και ε, προτεραιοτήτων, αλλά και ότι αυτέ οι προτεραιότητε που ορίζονται πράγματι εφαρμόζονται, πράγματι υλοποιούνται και πράγματι αξιοποιούνται τα χρήματα εκεί που θα έπρεπε. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι έχουμε όλοι συμφέρον και η Ρουμανία να παρουσιάσει σημαντικότερη πρόοδο στον τομέα αυτών. Περιμένω με αδειμονία πρέπει να πω να μου εντοπίσετε με την απάντησή σας πού βλέπετε ακριβώς τα προβλήματα, σε τι οφείλονται όλα αυτά. Κύριος Μπουστινάρου, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω ρουμανικά. Αναφέρω τη δήλωση του διοικητού ε, της Εθνικής Τραπεζής της Ρουμανίας ε, ότι οι πολιτικοί δείχνουν έτσι μια κομματική αντίληψη και μόνο. Η δυνατότητα από τη Ρουμανία απορρόφησης κονδυλίων είναι, ε, μας προκαλεί ανησυχίες. Εντάξει θα μπορούσε εδώ Μάλλον μόλις μάθαμε ότι η υπουργό ήρθε στο αεροδρόμιο του Ζαβεντέμ εδώ ξεκινώντας από τα συμπεράσματα της έκθεσης μας θα θέλαμε να έχουμε ε, μια καλή συνεργασία, είχα μια καλή συνεργασία με τα μέλη τη αντιπροσωπείας και τον κύριο Ρόι, τον πρόεδρο τη Επιτροπή. Θα ήθελα να υποβάλω ορισμένε ερωτήσει. Τι γίνεται με την περιφερειακή μεταρρύθμιση στη Ρουμανία. Αυτό ήταν από τα θέματα που μα απασχολούσαν, ήταν από τα σημεία κλειδιά τη εκθεσή μα. Δεύτερο, η ρουμανική κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξη τι κάνει για να βελτιώσει τι δυνατότητε, τι διοικητικέ και τι. Ε, και την αποτελεσματικότητα αυτής της και μετά από την έκθεση Σόρος. Τι γίνεται και το Ίδρυμα για μια ανοιχτή κοινωνία και η μελέτη η δικιά μου επίσης. Σε όλες αυτές τις αναφορές αναφέρεται μια ιδιαίτερα περισμένη διοικητική ικανότητα. Εδώ τι γίνεται στην ρουμανική διοίκηση, τι μπορεί να γίνει εκείνοι που διαχειρίζονται τα κονδύλια αυτά είναι ιδιαίτερα περισμένος ο αριθμός τους. Πώς, γιατί και επίσης υπάρξουν τα φορολογικά κίνητρα για τη χρησιμοποίηση αυτών των ε, κονδυλίων γιατί η κυβέρνηση ακύρωσε αυτά τα κίνητρα και επίσης ε, πριν από δύο εβδομάδες 2,2 ε, δισεκατομμύρια ευρώ πήραν ε, για την περίοδο μέχρι το 2014. Όλα αυτά τα ποσά για να μπορέσουν να αναπτύξουν ε, προγράμματα εκτός από την συγχρηματοδότηση την ευρωπαϊκή. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αυτά τα χρήματα δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με καλύτερο τρόπο για να αναπτυχθεί περισσότερη δυνατότητα ε, συγχρηματοδότησης και τι γίνεται με το ΦΠΑ και με την κρίση και δυστυχώς στη Ρουμανία η δυνατότητα συγχρηματοδότησης είναι ιδιαίτερα περισμένα. Θα ήταν πολύ καλύτερα όμως να ενισχυθεί αυτή η δυνατότητα συγχρηματοδότησης από πλευράς χώρας μου. Δεν θα ήταν καλύτερο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω τον κύριο Μοργιάνου για την παρουσία του για την παρουσίασή του επίσης βέβαια. Ακούσαμε πολλούς αριθμούς, πολλά ποσά, πολλά ποσοστά. Θα ήθελα όμως να επανέλθω στην ιδέα που ανέφερε ο κύριος Ρόι, ο συναδελφός μου. Εμείς γιατί μιλάμε. Μιλάμε για τον προϋπολογισμό από το 2014 μέχρι το 2020. Το κριτήριο απόδοσης και το επίπεδο απορρόφησης είναι πολύ σημαντικά σήμερα στη Ρουμανία είτε μας αρέσει αυτό είτε όχι είναι από τα κύρια στοιχεία και τις κύριες αντιρρήσεις των ευρωσκεπτικιστών ε, που είναι αντίθετη με την πολιτική σύνοχή για τη δυνατότητα να υπάρξουν τα ποσά αυτά στον προϋπολογισμό για τη συνοχή. Γιατί δυστυχώς η Ρουμανία δεν προσφέρει θετικά αποτελεσματά. Είναι το αρνητικό πρότυπο και ε, αν γίνει κάτι τέτοιο και η Ρουμανία θα χάσει, αλλά και όλοι μας θα χάσουμε και όλη η πολιτική συνοχή θα χάσει. Γι' αυτό θα πρέπει να δείξουν πόσο υπεύθυνη είναι από πλευρά ρουμανική κυβέρνηση. Επίση, μια συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί είμαστε διεθνή, σε διαρκή συνεργασία μαζί του και βλέπουμε ποιο θα πρέπει να είναι το πρόγραμμα δράση. Αυτό το πρόγραμμα δράση, από τη στιγμή που έχει εριστικοποιηθεί, τι γίνεται, εδώ γιατί μιλάμε, εδώ μιλάμε σε μια εξειδικευμένη ε, επιτροπή και δεν θα πρέπει να μιλάμε για γενικά πράγματα, θα μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες για τη Ρουμανία, τι γίνεται με αυτό το πρόγραμμα δράσης και εφαρμογή. γιατί αν αυτό το πρόγραμμα δεν εφαρμοστεί τάχιστα στη Ρουμανία και φτάσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου χωρίς να γίνει κάτι, θα είναι πολύ αργά. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα κύριε Μουρτζάνου να σας ρωτήσω το εξής. Πότε θα ξεκινήσετε με την εφαρμογή αυτού του προγράμματος δράσης. Και επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν το πρόγραμμα ε, δράσης αναφέρει και την επιστροφή του ΦΠΑ γιατί σίγουρα αυτό έχει να κάνει με τις τοπικές αρχές και με όλους ε, που θα ωφεληθούν από αυτή τη χρηματοδότηση. Ε, τι γίνεται με αυτή την επιστροφή του ΦΠΑ τι σχέση, πώς ε, ανακατεύονται και οι φορολογούμενοι, τι γίνεται με τα ε, συμβόλαια, με τις συμφωνίες που κλείνονται από πλευράς δημοσίου. Μήπως στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλα αυτά δεν θα πρέπει να ισχύσουν όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν σκεφτήκατε για μια απλοποίηση του ολοεγχειριδίου που ενημερώνει εκείνους που ζητούν αυτά τα χρήματα και ορισμένε απλοποίησει και την απάλληψη διαφόρων κριτηρίων που θίγουν την αποτελεσματικότητα και την καλή εφαρμογή αυτών των μέτρων και επίσης η κυβέρνησή σας και το Υπουργείο το οποίο εσείς εδώ εκπροσωπείτε είναι διατεθειμένο να αναγνωρίσει ότι χρειάζεται βοήθεια και να δεχτεί αυτή τη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια μιας τεχνικής αρρωγής ε, και με την ε, μετάβαση ορισμένων εμπειρογνωμόνων ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση όλων αυτών και για να βοηθήσουν τις ομάδες οι οποίες εργάζονται κάτω από την καθοδήγηση του Υπουργείου σας και γενικά της κυβέρνησης. Τι γίνεται με αυτή την τεχνική αρρωγή, αν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής όλων αυτών των προγραμμάτων που αναφέρουμε. Επίσης, ε, θα ήθελα να ακούσω τις απαντήσεις σας μετά από τις ερωτήσεις που μόλις σας υπέβαλα και επίσης θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο ακόμα. Εντάξει, εσείς και η κυρία Υπουργός και η κυβέρνηση σε τελευταίο λόγο ε, να καταλάβουν ότι δεν πρόκειται μόνο για προβλήματα της Ρωμανίας. Εδώ μιλάμε για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Θα ήθελα να επανέλθω στο σχόλιο του κυρίου Μπουστινάρου για τη συγχρηματοδότηση. Πέρα από τα 4,5 δισεκατομμύρια που πάνε στον προπολογισμό και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για την συγχρηματοδότηση και κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για το σκοπό αυτό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, οι προτεραιότητέ σας στα σχέδια αυτά, ποια είναι πριν από λίγο και μόνο καιρό εσείς ξεκινήσατε εγγενιάσοντες στο, σε αγροτικές περιοχές εγκαινιάσατε αθλητικές εγκαταστάσεις. Απ' την άλλη μεριά όμως εκεί δεν υπήρχαν σχολείο. Τι γίνεται, υπάρχουν προτεραιότητες ή κάνουμε ό,τι θέλουμε και ό,τι μας ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή σύμφωνα με τα συμφέροντά μας. Thank you, uh, Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον κύριο Υφυπουργό. Δυστυχώ εγώ δεν μπόρεσα να επισκεφθώ τη Ρουμανία στο τελευταίο ταξίδι, αλλά διάβασα την έκθεση και φυσικά συνομίλησα και με του συναδέλφου για διάφορα μελήματά του. Λυπούμε που μιλήσατε τόσο γρήγορα και ήταν δύσκολο να σα παρακολουθήσουμε ως αδύνατον. σω όμως μπορείτε να μας δώσετε κάποιε διευκρινήσεις τώρα με τι ερωτήσει. Είπατε πώ έχετε έναν εθνικό είπα το εκπρόσωπο. Καλή ιδέα μου φαίνεται αυτό. Νομίζω ότι είναι καλό. Κάποιος να βάζει τάξη όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Άρα κάποιος έχει διοριστεί, παρακολουθείτε και τις εξελίξεις και να λαμβάνει δράση αν χρειαστεί, αν υπάρξουν προβλήματα. Σε κάποια από τα αριθμητικά στοιχεία που κατέγραψα πάντως, βλέπω ότι από 11 δις ευρώ που έχουν ήδη δαπανηθεί, τα 4,6 εκατομμύρια πάνε στη διαχείριση κάτω από το 40% δηλαδή του συνολικού ποσού που δαπανάτε. Πάλι διορθώστε με αν κάνω λάθος τα νούμερα. Μου φαίνεται όμως πολύ υψηλό κόστος για διαχείριση, management. Και εγώ που προέρχομαι από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των φιλανθρωπικών οργανώσεων όπου έχουμε ε, πολλές φορές ε, χρησιμοποιήσει ε, δώρες Ξέρω πολύ καλά ότι σε κάθε καλό σχέδιο μπορεί κάποια στιγμή να διωγγωθούν πέραν του προβλεπωμένου τα, ε, το κόστος, να διωγγωθεί το κόστος διαχείρισης. Δεν κατάλαβα όμως από αυτά που είπατε αν ήταν σε εθνικό επίπεδο ή σε τοπικό το κόστος διαχείρισης τόσο υψηλό. Φανταζόμαι ότι η διαχείριση θα έπρεπε να ήταν σε πιο χαμηλό επίπεδο, δηλαδή εκεί που δαπανώνται πράγματι τα λεφτά. Ίσως μπορέσετε να, το διαχεί, να μας το διευκρινίσετε αυτό. Επίσης μας, είπατε, μας μιλήσατε για αιτήσιες συναντήσεις με την Επιτροπή για να υπάρχει παρακολούθηση των σχεδίων. Δεν νομίζω ότι αρκεί αυτή η συχνότητα. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχουν πιο συχνές ε, επαφές υψηλού επίπεδου μεταξύ της κυβέρνηση και της Επιτροπής για να υπάρξει παρακολούθηση αυτής της υλοποίησης. Και επίσης από αυτά που ακούμε από την έκθεση φαίνεται ότι οι άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν τα σχέδια χρειάζονται πιο πολύ υποστήριξη. και κατάρτιση, γιατί υπάρχει ανάγκη για ειδική κατάρτιση. Πρέπει κανεί να έχει ειδικέ γνώσει για να διαχειριστεί αυτά τα κονδύλια. Μερικέ φορέ λοιπόν. Αυτό που χρειάζεται για να βελτιωθεί η διαχείριση ενό προγράμματο, η υλοποίηση μάλλον ενό προγράμματο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά καλή κατάρτιση των ανθρώπων που καλούνται να το εφαρμόσουν. Πώ λοιπόν είναι εκεί το πρόβλημα. Έχετε δώσει κάποια έμφαση σε αυτό. Και κάτι ακόμη, και δεν έχω χρόνο. Πολλά φαίνεται είναι τα ποσά ευρωπαϊκών κονδυλίων που αποθηκεύονται σε τράπεζες της Ρουμανίας και ρωτώ, οι τόκοι αυτών των ποσών ξαναμπαίνουν στον Κορβανά ή χάνονται ή πηγαίνουν κάπου αλλού. Τι γίνονται αυτά τα χρήματα όταν δεν δαπανώνται όπω πρέπει. Η Πρόεδρο, αγαπητοί συνάδελφοι, οπως πρεπει η προεδρος αγαπητη συναδελφοι εχω κλεισει τον κατάλογο των αγορητών λόγω περιορισμού χρόνου και παρακαλώ όσοι είναι να λάβουν το λόγο να είναι στο δυνατόν πιο σύντομο. Ο κ. Σταυρακάκης, παρακαλώ. Uh, Κυρία Πρόεδρε και κύριε Μπουρτζιανάου, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ένας εκ των λόγων της χαμηλής απαρόφησης κονδυλίων είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι στα ευρωπαϊκά σχέδια. Δεν απασχολούνται αρκετοί άνθρωποι στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και αυτό αποδείχθηκε και από την επίσκεψή μας στη Ρουμανία τον Νοέμβριο. Όντως, ε, η πιο ε, οι η καλύτερη ε, υπάλληλοι θα προσελκυθούν από τι ε, υψηλέ αποδοχέ που να του προσφέρει ο ιδιωτικό τομέα. Μήπω θα έπρεπε λοιπόν ο δημόσιο τομέα να επανεξετάσει τι αποδοχέ των υπαλλήλων του σε κάποιο επίπεδο για να του κρατήσει. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υφυπουργέ, Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχά θα ήθελα να επισημάνω ότι ήμουν μέλος αντιπροσωπεία στη Ρουμανία και θα ήθελα να εκφράσω ρητέ ευχαριστίες προς τους συναδέλφους, Ρουμάνους τους συναδέλφους εδώ τη Επιτροπής, διότι μας ετοίμασαν ένα πρόγραμμα εξαιρετικό, με πολύ καλή επισκόπηση, ει βάθο μελέτη της κατάστασης περιφερειακή πολιτική στην Ρουμανία. Και είδαμε πολλά και συγκεκριμένα παραδείγματα. Αυτά που ανέφεραν λοιπόν, που εξέθεσαν μέχρι τώρα οι συνάδελφα και ιδιαίτερα ο κύριος Φανίστηλ Ρόι, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Η δική μου εντύπωση ήταν όντω, όπως και των συναδέλφων, ε, ότι ενώ περίμενα πως οι αρχές ε, της ε, τοπικής αυτοδιοίκησης όσοι είστε τουλάχιστον στη Γερμανία θα έριχναν όλα τα φταξίματα στις Βρυξέλλες και θα βρίζανε τις Βρυξέλλες συνέχεια ε, είδα ότι τι συμβαίνει αυτό είδα ότι μάλλον τα προβλήματα το πίσω στο επίπεδο της Ρουμανίας της ίδιας και επίσης η αυτοδιαχείριση των περιφερειών ή των κοινοτήτων φαίνεται ότι ακόμα δεν έχει προχωρήσει ε, με την ε, έμφαση που χρειαζόταν ε, σε επίπεδο περιφερειακής πολιτικής, πολιτικής συνοχής συγκεκριμένα. Γι' αυτό νομίζω θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και να κοιτάξουμε πού υπάρχουν ευθύνες στη φάση της υλοποίησης και να δουλέψουμε πάνω στις ευθύνες που θα εντοπιστούν. Δεύτερον, Επίση, ε, διαπίστωσα και είναι καλό αυτό για τη γερμανική οικονομία τουλάχιστον ότι πολλά από αυτά τα σχέδια τα έχουν αναλάβει να τα εκτελέσουν γερμανικέ εταιρείε. Τα έργα αυτά. Αλλά θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να παραλυφθεί διότι έχουμε και επανέρχομαι στο ίδιο σημείο σωστικά έχουμε να κάνουμε με πολλούς παράγοντες εμπλέκονται πολύ στη διαχείριση και στην εκτέλεση ενό έργου και τελικά το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα θέλαμε. Χάνεται πολύ χρόνο. Χρειάζεται βελτίωση λοιπόν στη διαχείριση. Πέραν των άλλων που αναφέρθηκαν. Και για άλλη μια φορά δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να συζητούμε μέσω, προ... συζητούμε μέσω πρόθεσμες δημοσιονομικές προοπτικές, στο μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο και βλέπουμε ότι ακόμα δεν έχει διασωθεί η πολιτική συνοχή. Ξέρουμε ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την αλληλεγγύη έτσι ώστε και τα κράτη που είναι καθαροί χορηγοί να στηρίζουν τα κράτη που έχουν κοινωνικές και άλλες αδυναμίες, διαφορετικές αδυναμίες, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται να αποδεικνύεται και ότι τα χρήματα αξιοποιούνται αποτελεσματικά. Εάν τα καταφέρουμε όλα αυτά μαζί, τότε όντως πιστεύω η πολιτική συνοχή θα έχει λαμπρό μέλλον. Ιδάλλως, η διαπίστωση θα είναι ότι δεν φέρνει το αναμενόμενο αποτέλεσμα πολιτική συνοχής, δεν κερδίζει η Ευρώπη χάρη στην πολιτική συνοχής και άρα Γι' αυτό θα ήθελα για άλλη μια φορά να απευθύνω την έκκληση προς τη Ρουμανία να ακολουθήσει το καλό παράδειγμα άλλων κρατών της πρόσφατης ένταξης που τα κατάφεραν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τα κονδύλια της τελευταίας περίοδου και να τα αξιοποιήσουν εκεί πραγματικά υπήρχε ανάγκη. Ευχαριστώ κύριο Σμότουλο a vrea i eu să... ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστώ Για άλλη μια φορά, για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε αυτή η επίσκεψη της αντιπροσωπείας. Και να ευχαριστήσω για την υποδειγματική συνεργασία με τους συναδέλφους των άλλων ομάδων με την ευκαιρία αυτή. Εμεί, οι Ρουμάνοι συνάδελφοι τουλάχιστον οργανώσαμε από κοινού την επίσκεψη και προσπαθήσαμε μέσα από αυτή την επίσκεψη, μέσα από το ταξίδι να αξιοποιήσουμε όσο μπορούσαμε και την εμπειρία τη ιδιαίτερη γνώση που έχουν οι άλλοι συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φερρυπίν, επιτάχυνση της ε, ροής των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ναι, υπάρχει αδύρυτη ανάγκη στη Ρουμανία να βελτιωθούν, να βελτιωθούν αυτές οι επιδόσεις όπως βλέπουμε ότι υπάρχει αντίστοιχα ανάγκη και σε άλλα καινούργια σχετικά κράτη-μέλη. Θα πρέπει, και θα ήθελα να το πω αυτό ε, ξεκάθαρα, να επιταχύνουμε την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και ένα έγγραφο υποσυζήτηση αυτή τη στιγμή, ένα έγγραφο εργασίας του συναδέλφου Τόιρερ που έχει να κάνει με την απορρόφηση των κονδυλίων από το Διευθυντικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όπου αναφέρεται στην περίοδο 2007-2013 σε πληρωμές και στα κράτη που πρόσφατα εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατάσταση παρουσιάζεται ως εξή. Στην απορρόφηση 11% Βουλγαρία, 14% Ρουμανία, Ελλάδα 16%, Πορτογαλία 17% στα πρόσφατα μέλη, 19% η Τσεχία και 20% η Πολωνία. Άρα, αναλογικά η Ρουμανία δεν απέχει πολύ από το μέσο όρο Τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι στο 21%. Αλλά βέβαια θα πρέπει να επιταχύνουμε τους ρυθμούς μας, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και ίσως θα ήταν καλό να καθοδηγηθούμε και από καλές πρακτικές που έχουν αναπτύξει άλλα κράτη-μέλη. Επίσης, θα θέλαμε να ε, αναπτυχθούν περισσότερο οι βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των ρουμανικών περιφερειών. Δηλαδή, εκεί όπου βλέπουμε, όπως είπε και ο κύριος Μποσινάρου νωρίτερα, καλές ε, επιδόσεις, η δυτική περιφέρεια Φερρυπίνη της Ρουμανίας, όπως αναφέρθηκε, που είδαμε στην επίσκεψή μας, θα μπορούσε να αποτελέσει έμπνευση και για τις υπόλοιπες ε, περιφέρειες. Ξέρουμε τώρα ότι έχει κάνει προσπάθειες το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ρουμανίας. Έχει τους τελευταίους ε, έξι μήνες απορροφήσει κονδύλια το, ισοδύναμα με αυτό των τελευταίων 6,5 ετών. Φυσικά πάλι δεν αρκεί αυτό και πάλι χρειάζεται επιτάχυνση των ρυθμών. Ε, διαφορετικά θα τα καταφέρει η Ρουμανία όπως θα έπρεπε. Και γι' αυτό θα ήθελα να καταλήξω τώρα, γιατί δεν έχω χρόνο, για να απευθύνω έκκληση για άλλη μια φορά για έναν για ένα πρόβλημα, διότι ναι χρειάζεται τα κονδύλια αυτά, η Ρουμανία, χρειάζεται όμως ταυτόχρονα και προγράμματα που θα αναπτυχθούν στο εσωτερικό της χώρας, από το δικό της τον προπολογισμό δηλαδή. Δηλαδή, πέραν της συγχρηματοδότησης που τους άλλους προβλέπεται για τα ευρωπαϊκά προβλήματα, προγράμματα, θα πρέπει η Ρουμανία να αναπτύξει και δικά της προγράμματα από τον εθνικό της προπολογισμό. Μάλιστα εδώ σε μια διπλανή αίθουσα ε, που έγινε μια εκδήλωση για τα 20 χρόνια της επανένωσης της Ευρώπης και έρθει ο Ζακ Ντελόρο είδους και είπε ότι 140 δισεκατομμύρια ευρώ επένδυσε ή μάλλον δια, ε, μεταβίβασε Δυτική Γερμανία στην Ανατολική την εποχή της Επανένωσης και πάλι αυτά δεν ε, αποδείχθησαν επαρκή για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες και οι καθυστέρηση στην ανάπτυξη. Ε, τέτοια κονδύλια χρειάζεται η Ρουμανία, χρειάζεται λοιπόν και την υποστήριξη απ' έξω, αλλά χρειάζεται και δικά της κονδύλια, χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται σκληρή δουλειά και πιστεύω χρειάζεται και σε αυτό χρειαζόμαστε βοήθεια από εσά, τεχνογνωσία, know-how εξειδίκευση, ειδικέ γνώσεις που πιστεύω μπορείτε να μας προσφέρετε εσείς οι συνάδελφοι από τα άλλα κράτη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Λούχαν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστώ και πάλι τον, και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Υφυπουργό. Ήταν πολύ ε, οι πληροφορίες που μας έδωσε, διεξοδικές. Βλέπουμε βέβαια ότι η ρουμανική κυβέρνηση έχει κάνει πολύ σκληρή δουλειά. Την ευχαριστούμε. Και χρειάζεται, πιστεύω, μια ουσιαστική εφαρμογή της πολιτικής της ε, συνοχής στη Ρουμανία. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε για το επόμενο δημοσιονομικό πρόγραμμα 2014-2020 τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Για την περιφερική ανάπτυξη έχουμε ακόμα ένα σχόλιο που δεν ανέφερε ο Υφυπουργό και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Το Υπουργείο έχει 2, έχει 2,6 φορές παραπάνω σχέδια από ό,τι τα χρήματα που διαθέτει. Άρα λοιπόν το Υπουργείο έκανε δουλειά του. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ειδικά προγράμματα εφαρμογής αυτής της πολιτικής στη Ρουμανία. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι η πολιτική περιφερικής ανάπτυξης. Νομίζουμε ότι σε άλλα πλαίσια αντιμετωπίζει προβλήματα η Ρουμανία. Εάν πάρουμε υπόψη μα όμω τα χρήματα που πάνε στη τέσσερα πρώτα χρόνια στη Ρουμανία, η δυνατότητα απορρόφησης της Ρουμανίας είναι πάνω από 18%. Μέσο όρο ο ευρωπαϊκό είναι 21%. Όχι, άρα λοιπόν δεν είναι το κακό παράδειγμα. Είμαστε λίγο παρακάτω από το μέσο όρο απορρόφηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι τα κύρια στοιχεία τα οποία χρειάζεται εδώ να αναλύσουμε για να βελτιώσουμε την πολιτική συνοχή είναι διαφορετικά θα πρέπει να δούμε ας πούμε την πολυδιαχείριση ένα στοιχείο που τώρα τελευταία υποστηρίχθηκε από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως επίσης η βελτίωση της χρησιμοποίησης. Θα πρέπει να δούμε όμως ότι και άλλες χώρες πέρασαν από τον ίδιο δρόμο με τη Ρουμανία μια εκμάθηση τα του τι πρέπει να κάνουν στην αρχή. Θα πρέπει να θυμηθούμε για την ένταξη της ε, την, ε, για την ένταξη της Ρουμανίας ότι υπήρξαν ήδη καθυστερήσεις από την κυβέρνηση Ρουμανίας ε, και απαιτήθηκε τουλάχιστον ένα έτο για να συνταχθεί ο οδηγό για τη χρησιμοποίηση αυτών των στοιχείων, αυτών των κονδυλίων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θα μπορούσε να συνταχθεί νωρίτερα. Γιατί δεν έγινε, εντάξει. Τώρα είναι εύκολο να επιτίθεται κανεί στην κυβέρνηση αυτή από τη στιγμή που άλλοι δεν έκαναν το καθήκον του παλιότερα. Εμεί θα πρέπει να δούμε τη δυνατότητα ακριβώ εφαρμογή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμογή όλων αυτών των σχεδίων. Νομίζω ότι είναι ανωδική η τάση, όπως είπε συνάδελφος Μαξούλα, ότι την τελευταία χρονιά η δυνατότητα ήταν ε, σε το σύνολο των τριών προηγουμένων ακόμα ετών. Άρα λοιπόν υπάρχει μια γεωμετρική αύξηση και ανάπτυξη και δυνατότητα απορρόφησης. Είμαι αισιόδοξο και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να περβούμε στο τέλος περίοδο το 90%. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω από τον Υφυπουργό να απαντήσει και να σχολιάσει. Ακούστηκαν πολλά, πολλά ερωτήματα και πολλές ανησυχίες. Γνωρίζουμε ότι η Ρουμανία πρέπει να εξυγχρονίσει την οικονομία και την κοινωνία. Υπάρχει υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά θα θέλαμε να απορροφάτε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Υπήρχαν πολλές συστάσεις ε, από τους συναδέλφους, πολύ λεπτομερείς ερωτήσεις, ε, αλλά υπήρχε και μια γενική συνένευση γύρω από την διοικητική ε, υποδομή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν να μας απαντήσετε στα σχόλιά μας αυτά και να μας ε, διαβεβαιώσετε ότι η ρουμανική κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να επενδύσει όσο το δυνατόν καλύτερα και όσο το δυνατόν συντομότερα την ε, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ναι, σας ευχαριστώ γιατί η δυνατότητα απορρόφησης ήταν τόσο χαμηλή. Αυτό ρωτήθηκε. Αλλά σας λέω ότι το 2007 αυτό που σχεδιάστηκε το σεβόμαστε. Το πρόβλημα ποιο είναι. Είμαστε κάπως διστακτικοί γιατί υπάρχουν αφιβολίες όσον αφορά την ικανότητα εκείνων που θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα κονδύλια για να εφαρμόσουν αυτά τα σχέδια. Αυτά λοιπόν και ακόμα το κύριο πρόβλημα που έχουμε με εκείνους που παίρνουν αυτά τα χρήματα είναι ότι όσοι εργάζονται για τα κοινοτικά προγράμματα δεν πληρώνονται καλά. Ε, γιατί αν εργάζονται καλά πάνε στον ιδιωτικό τομέα που πληρώνονται καλύτερα είτε περνάνε σε άλλες δραστηριότητες όπου επαναλαμβάνω οι αμοιβέ είναι υψηλότερε. Για να επιστρέψουμε τώρα σε αυτό που έλεγε ο κ. Μποστινάρου να σας πω ότι εμείς ε, δεν που κάναμε ε, παλιότερα και τώρα η δημόσια διοίκηση πληρώνει μέχρι και 75% παραπάνω αμοιβέ σε αυτούς τους διαχειριστές. Αυτό το διέταξε το ρυθμισή κυβέρνηση από την αρχή του χρόνου και όλοι όσοι εργάζονται για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και η τοπική διοίκηση έχει πρόσβαση στις σχετικές εκτιμήσεις και μπορεί και να πληρωθεί όπως είπαμε μέχρι και 75% παραπάνω να αμοιβθεί και θα πρέπει να δούμε και τι να τα από τα κονδύλια κονδύλια αυτά, γιατί δεν είναι όμω σωστά, γιατί τελικά θα είχαμε λιγότερα σχέδια που θα εγκριθούν, άρα λοιπόν καλύτερα από τον δικό τους προϋπολογισμό να πληρώνονται, από τον δημόσιο προϋπολογισμό. Τώρα, η παριθμόν 69 ε, αρρύθμιση της κυβέρνησης επιτρέπει στις τοπικές αρχές για την συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων να δανείσουν χρήματα πάνω από το όριο που καθορίζεται από τον νόμο. Επιπλέον δηλαδή ένα 20%. Έτσι οι τοπικές αρχές μπορούν να ρυθμίσουν καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά τα προβλήματα τα οικονομικά. Για τα μέτρα τώρα που διαθέτουμε, εντάξει, να σας πω εδώ το πρόγραμμα αυτό δεν είναι πλήρες. Θα το δούμε, θα είναι περίπου στις 15 Απριλίου θα ολοκληρωθεί. Θα σας το αποστείλω αυτό το έγγραφο έτσι όπως το έχουμε τώρα. Πρόκειται για μια χρήσιμη πληροφορία για σας. Είναι δημόσιο το κείμενο αυτό, δεν είναι απόρριτο, δεν είναι εμπιστευτικό, δεν θέλω να σας το κρύψω και θα δείτε εδώ απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που υποβάλλατε. σχετικά με το ΦΠΑ. Το 2009 ξεκινήσαμε μια διαδικασία με τις τοπικές αρχές. Τι έγινε όπως το γνωρίζετε, τα τιμολόγια, οι αποδείξεις ε, ε, βγαίνουν στις τοπικές αρχές και εμείς θα πρέπει να τα εγκρίνουμε. Έχουμε ένα 15% περιθώριο που απομένει στο, στις τοπικές αρχές να το πληρώσουν από τη στιγμή που θα έχουν τα χρήματα για να πληρώσουν όλα τα έξοδα. Επιπλέον λοιπόν ένα περιθώριο 15%. Όταν πρέπει να πληρώσουν το ΦΠΑ, δεν θα πρέπει αυτός να ενταχθεί στον τοπικό προπλησμό. Αυτό μέχρι το 2009 πληρώναμε 15% προκαταβολικά για τις εργασίες και 15% για φορισμένους συμβούλους, διαβουλεύσεις κλπ. Τώρα, για τις τράπεζες Να σας πω για τα επιτόκια. Τι πληρώνεται για τα χρήματα που είναι στραπέζες. Όλοι αυτοί οι τόκοι πάνε στη χρηματοδότηση των σχεδίων και αυτό σε μηνιαία βάση γίνεται και Πού πάνε, όπως είπα, στη χρηματοδότηση αυτών των σχεδίων. Είναι μια απόλυτα διάφανη διαδικασία. Επίσης αναφερθήκατε στις δημόσιους διαγωνισμούς, δημόσιες ε, συμφωνίες του δημοσίου και αναγνωρίζω ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που θα πρέπει να ρυθμιστεί στο μέλλον σχετικά με αυτά που ανατίθενται από το δημόσιο και χρειάζεται να ξεκινήσω από μια αφετηρία ότι εμείς ε, βέβαια δεν είμαστε εκείνοι που οργανώνουμε αυτούς τους πλειοδοτικούς ή μοδοτικούς διαγωνισμούς ε, θα πρέπει να δούμε ότι όλα αυτά γίνονται σε επίπεδο τοπικής διοίκησης. Ε, εντάξει, μπορούμε να ασκήσουμε ένα έλεγχο μόνο εάν υποψιαζόμαστε κάτι. Ε, αν υποψιαζόμαστε τότε στέλνουμε μια επιστολή στις δύο δημόσιες αρχές που προχωρούν σε αυτή την επαλήθευση, στον έλεγχο, γιατί εμείς στο Υπουργείο δεν έχουμε το απαραίτητο μέσο για να προβούμε στο σχετικό έλεγχο. Εάν όμως κάτι υποψιαζόμαστε, όπως είπα, τότε το ανακοινώνουμε αυτό στις δύο αρχές οι οποίες είναι οργανωμένες για αυτόν τον έλεγχο και δυστυχώς υπάρχουν αρκετά προβλήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Σχετικά τώρα με τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την βοήθεια που μπορεί να μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το κάνουμε. Έχουμε το Ζάσπερα, ας πούμε. Έχουμε μια τεχνική αρρωγή και τους στείλαμε ήδη σχέδια για να τα ελέγξουν εκείνοι και να επαληθεύσουν. Όχι ότι έχουμε, τρέφουμε αμφιβολίες και υποψίες ότι έχουμε, αλλά είναι με πολλά χρήματα σχέδια, προγράμματα. Αυτό καλύτερα να κάνουμε ένα πλήρη έλεγχο μέσω του και εμείς εργανόμαστε συνεχώς ε, προς αυτή την κατεύθυνση και μιλάω για το επιχειρησιακό τοπικό πρόγραμμα, όχι για άλλα σχέδια. Εμείς επαναλαμβάνω, συνεχώς είμαστε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον έλεγχο όλων αυτών. Η κυρία Μανέσκου επίσης ρώτησε κάτι, ρώτησε κάτι σχετικά με το εγχειρίδιο για τον χρήστη. Εκεί επιφέραμε αρκετές μεταβολές, αλλαγές και δεν μπορούμε όμως να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο γιατί τότε θα πρέπει να έχουμε ένα καινούριο έλεγχο, ένα έλεγχο που ήδη πραγματοποιήσαμε το 2007-2008 τον είχαμε διεξάγει αυτόν τον έλεγχο και χρειάζεται να τα δούμε όλα αυτά, να δούμε τι μπορούμε να ρυθμίσουμε, τι μπορούμε να αλλάξουμε δρόμο κάνοντας. Και εδώ θα πρέπει να δούμε και του συμβασμού του πολιτικούς, το ένα το άλλο δεν θέλω να μπούμε τώρα σε τέτοιου δρόμους εμείς. Πάντως όλοι οι χρήστες συμφωνούν με όσα γίνονται και με τη θέση την οποία μέχρι τώρα υιοθετήσαμε. Τώρα σχετικά με τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, είναι δικέ πληροφορίε. Εμεί δεν έχουμε καμία πληροφορία προ την κατεύθυνση αυτή. Δεν ξέρω εσεί γιατί, σε τι πράγμα αναφέρεστε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό για τα 4,5 δισεκατομμύρια. Ναι, ακούστε, ακούστε, είναι κονδύλια τα οποία προσφέρονται στους Δήμους για σχέδια, ας πούμε, υποδομών, για αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλα σχέδια. Είναι τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ και σημαίνει ότι η δυνατότητα χρηματοδότηση είναι ακόμα χαμηλότερη. Τι γίνεται είναι το εθνικό πλαίσιο ε, χρησιμοποίησης αυτό, επένδυσης. Δεν είχα καταλάβει σε τι αναφέρεστε. Εντάξει, θα μπορούσα να σας πω μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, δεν πήραμε στα χέρια μας χρήματα. Αυτά είναι εικονικά χρήματα. Το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων είναι το εξής. Τι γίνεται συντάσσουμε ένα κατάλογο με προγράμματα ξεκινώντας ε, εντάξει υποδομής, ε, μεταφορών, ε, είτε προγράμματα για αποχετεύσεις, για παροχή πόσιμου ύδατος και για τα για τις διάφορες συμφωνίες θα πρέπει να έχετε και ιδιωτικές επενδύσεις γιατί δεν σας δίνει τίποτα ο δημόσιος προϋπολογισμός. Το 2009 όταν κλείσαμε αυτόν τον κατάλογο είδαμε ότι είχαμε πάνω από 13 δισεκατομμύρια προγράμματα ενώ στην αρχή είχαμε ξεκινήσει με 5 δισεκατομμύρια είχαμε σχέδια, τα προγράμματα που μέσω του Εθνικού Προγράμματος Επενδύσεων δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν. Τότε ξεκινήσαμε μία συζήτηση, μία ανάλυση στα πλαίσια του Υπουργείου μας και είπαμε ότι για όλα αυτά τα προγράμματα που έχουν υποβληθεί ε, ξόδεψε πολλά χρήματα ο κόσμος για να δει αν όλα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν, να πραγματοποιηθούν και θα πάνε χαμένα αυτά τα χρήματα. Είναι κρίμα έστω και αξιόλογα αν ήταν αυτά τα προγράμματα να μην εφαρμοστούν, να μην πραγματοποιηθούν. Θα ήταν κρίμα αλλά ίσως σε 4-5 χρόνια θα αλλάξουν ταυτόχρονα όμως και τα τεχνικά, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι τεχνικές απαιτήσει. Και τότε το 2009 είπαμε ότι οι πρώτες επενδύσεις που γίνονται γίνονται βάσει του δεύτερου άξονα, του δεύτερου προγράμματος αυτού και είπαμε στη συνέχεια ότι αυτό που παραμένει στο 312 στη Γεωργία ας πούμε οι δήμοι εκείνοι που δεν θα είχαν την απαραίτητη χρηματοδότηση και εκείνοι οι δήμοι όμως χρειαζόταν χρήματα και μπήκαν στα πλαίσια του εθνικού, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος επενδύσεων. Η δική μας η λογική, δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο, δεν είμαστε άμεσα ανανεμειγμένοι σε αυτό το εθνικό πρόγραμμα επενδύσεων, αλλά η λογική η γενική ήταν αυτή. Σχετικά λοιπόν με, την, ε, με τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Εντάξει, εύκολο ήταν ε, να καταλάβω τη θέση των δημάρχων στις τοπικές αρχές και να καταλάβω ποια τι αποτελούσε εμπόδιο. Και αυτό ακριβώς προχωρήσαμε σε μεταβολές, σε αλλαγές στον οδηγό του χρήστη. Να σας προσφέρω ένα σύντομο παράδειγμα. Ένα ένας δήμαρχος ήθελε ας πούμε να φτιάξει ένα αγωγό ε, δίπλα σε μια συνδρομική οδό δεν μπορούσε να το κάνει γιατί υπήρχε κάτω από το γεφύρι ας πούμε ε, μια στήριξη που ήταν δικαιοδοσία του Υπουργείου Μεταφορών. Άρα λοιπόν δεν μπορούσαμε να βάλουμε χέρι εμείς. Και ζητήσαμε την άδεια ε, να παρέμβουμε έστω και αν ήταν σε απογορευμένη, προστατευμένη ας το πούμε έτσι για μας περιοχή και το κάναμε αυτό σε πολλά προγράμματα μέσω των μεταβολών αυτών έγιναν πολλές παραχωρήσεις, έγιναν πολλά θετικά πράγματα ακριβώς επειδή εμείς θελήσαμε να έχουμε μια γενική εικόνα και όχι μόνο αυτό που κάνει ένα και μόνο Υπουργείο στενή οπτική δηλαδή δεν ξέρω αν υπήρξαν άλλες ερωτήσεις αν είναι ναι, ναι. μια ερώτηση για την περιφερειακή μεταρρύθμιση. Θα ήθελα εδώ να κάνω ένα προσωπική φύσεως σχόλιο πέρα τώρα από το τι φρονεί πολιτικά ο καθένας. Εδώ πρόκειται για μια βούληση πραγματική πολιτική. Θα θέλουμε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή λύση στην όλη αυτή διαδικασία ε, περιφερικής αντομετώπισης θετικής της χώρας. Εντάξει, και είναι και δική μου προσωπική άποψη αυτή οι περιφέρειες ε, οι ρουμάνικες δεν έχουν νομική υπόσταση γιατί αν το είχαν αυτό μέσω ενός κυβερνήτη, ενός περιφερειάρχη δεν ξέρω τι, τότε οι αρχές αυτές θα μπορούσαν να πάρουν άμεσα τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να περάσουν από ένα εθνικό Υπουργείο. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε στο μέλλον λοιπόν. Εδώ γιατί πρόκειται. Πρόκειται για επίδειξη πολιτικής βούλησης. Χρειάζεται να το συζητήσουμε στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο και χρειάζεται να πετύχουμε να βρούμε μια λύση. Ο ρόλος του Υπουργείου είναι να μπορέσει να απτύξει ομοιόμορφα την Ρουμανία να υπάρξει μια καλή συνοχή κλπ. Παραλαμβάνω όλα αυτά είναι δική μου προσωπική άποψη τίποτα περισσότερο. Δεν ξέρω αν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας. Διαφορετικά εντάξει, αν θέλετε να απαντήσω και σε άλλα, αν μου τα υπενθυμίσετε. Εδώ θα σας αφήσω το πρόγραμμα δράσης που διαθέτουμε για να το, διαβάσουν, ε, για να το διαβάσετε εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φεπουργέ. Εκ μέρου όλων των συναδέλφων ήταν ε, πάρα πολύ χρήσιμη η ανταλλαγή ε, απόψεων. Επίσης ε, θα θέλαμε να λάβετε και το μήνυμα ότι ελπίζουμε να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος σε σχέση με την απορρόφηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στη Ρουμανία και ελπίζουμε επίσης ότι αυτή η πιο συνετή απορρόφηση θα επισπευθεί γιατί θέλουμε η Ρουμανία να αποδείξει ότι η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντική για τις χώρες ε, που ε, πρέπει να προλάβουν τις υπόλοιπες και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώνεται η οικονομία τους και η αγωνιστικότητά τους. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ μία ακόμη φορά θα συνεχίσουμε με τη συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα περάσουμε στην ψηφοφορία, οπότε ας ελέγξουμε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες και κατά πόσο δουλεύει το σύστημα. Μπορούμε να αρχίσουμε την ψηφοφορία. «35 κάρτες» βλέπω εγώ από τις 36. Βλέπω όμως ότι είναι πολύ περισσότεροι στην αίθουσα. Μπορείτε παρακαλώ όλοι να βάλετε τις κάρτες σας στα μηχανήματα για να μπορέσουμε να ελέγξουμε αν δουλεύουν όλα τα μηχανήματα. Ωραία, περνάμε στην πρώτη ψηφοφορία. Έχουμε πέντε ψηφοφορίες στο σύνολο, αρκετά μακροσκελής. Πρώτον, Σαμπίν φερχέιν για τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα βριζονικότητας. Αρχίζουμε με τη συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7 απο, αποσύρεται. Περνάμε στη συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά τμήματα ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται καλύτερα να γίνει όμως ηλεκτρονικός έλεγχος της 23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 κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 59 άρχεται η ψηφοφορία Από το ΕΛΚ ψήφισε ένας παραπάνω. Μπορεί κάποιος να μην ψηφίσει. Δεν ξέρω πώς θέλετε να το κάνουμε. Αλλά πέρας ψηφοφορίας. 30 υπέρ 12 κατά. Εγκρίνεται. Ωραία. Συνολική ψηφοφορία υπέρ. Κατά. Α, ηλεκτρονικός πρέπει να ψηφίσουμε. Συγγνώμη, μα δεν το έχω γραμμένο, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικό στο τελικό κείμενο. Πέρα της ψηφοφορίας. 38 υπέρ και μία ψήφος κατά. Περνάμε στην ε, δεύτερη μας ψηφοφορία. Λουίς Παύλο Άλβες για τις κοινωνικές υπηρεσίες ε, κοινής ωφελίας. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος της ε, τροπολογίας 4. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος της 9. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στη συμβιβαστική 3. Διορθώνει η πρόεδρος. Ξέχασα τη 10. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 αποσύρεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 37 υπέρ, 4 ψήφοι κατά. Συγχαρητήρια στον Λουίς Παόλο Άλβες. Περνάμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Σεκέρσκι για την ε, κοινή γεωργική πολιτική μέχρι το 2020. Συμβαστική 1. Υπέρ. Ναι, παρακαλώ κύριε Κρέλ. Μία παρατήρηση μόνο για το παράδειγμα αυτό, επί τη ευκαιρία αυτού του παραδείγματο. Ψηφίζουμε τροπολογίε ε, οι οποίε δεν έχουν καμία σχέση με την περιφερειακή πολιτική, αλλά αποκλειστικά με τη γεωργία. Θα έπρεπε και οι γραμματεία αλλά και οι συνάδελφοι στο μέλλον να μεριμνούν έτσι ώστε να κοιτάμε θέματα τα οποία είναι δική μα αρμοδιότητα. Εγώ αισθάνομαι τύψει όταν είμαι υποχρεωμένη να καταψηφίζω ή να απέχω σε πράγματα ή να εγκρίνω πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω, γιατί δεν είναι της ειδικότητάς μου. Σημειώνουμε την παρατήρηση. Σημειώνουμε την παρατήρηση αυτή. Ούτω ή άλλω είχαμε και μια συζήτηση για την ε, γνωμοδότηση αυτή. Οπότε ε, το είχαμε αναφέρει και τότε. Πάντω είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε για το μέλλον. Πρέπει όμω τώρα να ψηφίσουμε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 Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικό στη 36. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ο κύριος Βλάσακ ε, έχει μία προφορική τροπολογία για την 45. Η 42 έχει αποσυρθεί. Α, συγγνώμη. Προφορική τροπολογία του κυρίου Βλάσακ για την τροπολογία 45. Θα ήθελα κυρία Πρόεδρε να σας πω ότι θα ήθελα στο τέλος της τροπολογίας αυτής μετά από την κλιματική αλλαγή και την καινοτομία να αλλάξουμε ως εξή, συμπεριλαμβάνοντας τον εξυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση της γεωργίας και της εκπαίδευσης. Διαφωνεί κανείς με την τροπολογία αυτή την προφορική? Αν όχι, οπότε ψηφίζουμε όπως τροποποιήθηκε. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 49 έναρξη ψηφοφορίας πέρας εγκρίνεται Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58. Υπέρ. Καταπίπτει 58. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 καταπίπτει 63 υπέρ κατά έλεγχος της 63 έναρξη ψηφοφορίας απορρίπτεται κατά πολύ Οπότε πάμε στην 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64 καταπέπτει. Καταπίπτει οπότε στην 60, 65. 66. Ψηφίζουμε την 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην 70. Υπέρ κατά αποχές έλεγχος της 70 έναρξη ψηφοφορίας Ψηφίζουμε λοιπόν την 70 έναρξη ψηφοφορίας Πέρας εγκρίνεται Η κυρία Κρόιλ. Ενδεχομένω να έκανα λάθο, αλλά νόμιζα ότι εφόσον εγκρίναμε την 62, άρα τότε δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε την 66 και την 67. Και την ψηφίσαμε, τι ψηφίσαμε. Θα ακυρώσουμε τότε τις ε, ψηφοφορίες που δεν χρειάζονταν. Πάμε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 Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το συνολικό κείμενο του σχεδίου γνωμοδότησης. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Περνάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία της γνωμοδότησης του κυρίου Τσέλερ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα παρακαλέσω τους συντονιστές να δώσουν λίγο προσοχή και να μου πούνε εάν μπορούμε να ψηφίσουμε on block τις συμβαστικές. Κυρία Σρέντερ, όχι. Μια γενική παρατήρηση, Πρόεδρε. με ενοχλεί το γεγονός ότι υπάρχει μια παρουσίαση εδώ στον, στον καταλόγο των ψηφοφοριών μας σαν να πρόκειται να ψηφίσουμε on block ενώ δεν μας έχει ρωτήσει κανείς. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι θα πρέπει αυτό να συμβαίνει μόνο όταν και εφόσον έχουν συμφωνήσει προκαταβολικά όλες οι ομάδες χωρίς καμία διαφωνία. Και πρέπει τότε ο κατάλογο του ψηφοφοριών να διαμορφώνεται κατά τρόπο να μπορούμε να τον επαληθεύσουμε, ώστε να μην υπάρξει κανένα λάθο, να μην παρισφρήσει κανένα λάθο, πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί αυτή τη στιγμή από πλευρά τη Γραμματεία. Δεν υπάρχει συμφωνία λοιπόν. Και παρακαλώ, οι συμβαστικέ αλλά και αντίστοιχε ε, τροπολογίε, αυτέ που καλύπτονται δηλαδή από το συμβασμό, να παρουσιάζονται έτσι ώστε να είμαστε θέση να κάνουμε την ψηφοφορία σωστά και με βάση τους κανονισμούς μας, αλλά και τώρα μεν μπορώ να δεχθώ να γίνει ψηφοφορία όπως προτείνεται, αν συμφωνούν οι λοιπές ομάδες, αλλά παρακαλώ στο μέλλον να μην επαναληφθεί αυτό. Και να έχουμε ένα πιο καθαρό κατάλογο ψηφοφοριών. Και επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι θέλαμε να ψηφίσουμε χωριστά την 4 και 10 συμβαστικές τροπολογίες. Η πρόεδρος. Καλώς. Ε,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 αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά ας επαληθεύσουμε για τη 18 παρακαλώ άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται η 20 τώρα σε τμήματα Πρώτο τμήμα της 20 υπέρ, κατά αποχές το Δεύτερο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 25 ε, τώρα, 25 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται, Κάθριν. Μα δεν ψηφίσαμε τη 19, πρόεδρε. Το συγγνώμη, κάποιο το τηλέφωνο έχει μείνει αναμένο και δημιουργεί παράσιτα. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 έχει αποσυρθεί, 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά. Νομίζω ότι είχε απορριφθεί, αλλά στην επαληθεύσουμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία απορρίπτεται. Στην 60. Παρακαλώ, κύριε Ρο. Χωρίς μικρόφωνο, μιλτής δεν ακούγεται. Παρακαλώ, μήπως θα μπορούσατε να ανοίξετε το μικρόφωνο σας ή τα δίπλα της κυρίας Ντελή, κάποιοι τέλος πάντων. Εντάξει, λειτουργεί. Θα δούμε, θα δούμε. 67 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε την 67. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασμα. Ε, συγγνώμη, αλλά δεν πρόλαβα να δω το αποτέλεσμα. 29 κατά. Α, υπέρ, υπέρ. Εγκρίνεται. Η 67 πάμε στην 69 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ. Όχι, σε παληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Ας κάνουμε την ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Έχει προφανώς εγκριθεί και σας ευχαριστώ, συγχαρητήρια. Και τώρα, τελευταία ψηφοφορία. Γνωμοδότηση Χίμπνερ, αν δεν κάνω λάθος, είναι η τελευταία. Θέλει κανείς το λόγο. Πάλι ρωτώ αν μπορούμε να ψηφίσουμε ε, ομαδών της ε, προτάσεις. Είναι έξι συνολικά. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Καλώς λοιπόν ψηφίσουμε τις τροπολογίες υπαριθμών 1 έως και 6 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τη λογική σκέψη 7 παρακαλώ. Μάλλον τροπολογία 7 κατά αποχές συνολική Ψηφοφορία ηλεκτρονική τώρα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στο σχέδιο έκθεση του κυρίου Βλασάκ, πρόγραμμα για το Ευρωπαϊκό Αστικό Περιβάλλον και το μέλλον του στο πλαίσιο τη πολιτική συνοχή. Να πάρει το λόγο, παρακαλώ, εσεί, δεν είστε έτοιμοι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω προσφέροντάς σας διάφορες πληροφορίες για την έκθεση αυτή για την πολιτική της συνοχής και το πρόγραμμα για το ευρωπαϊκό αστικό περιβάλλον. Θα πρέπει να δούμε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ε, η έκθεση αυτή δείχνει διάφορες εξελίξεις ε, τωρινές που τις παρατηρήσαμε ακριβώς την τελευταία περίοδο προγραμματισμού. Εδώ ασχολούμεθα με τις πόλεις και το ρόλο του στην πολιτική συνοχής. Θα ήθελα όμως να σας πω στην εισαγωγή ότι τώρα που θα πρέπει να προσφέρουμε χρήματα κοινοτικά θα πρέπει να δούμε τι είναι αγροτικές περιοχές, να υπάρξει μια συνδυασμένη ανάπτυξη και των αστικών περιοχών όμως και των, και των αγροτικών περιοχών. Επίσης να τονίσω τρεις ε, τροπολογίες για τις ε, για την κοινή πολιτική που υιοθετήσαμε πριν από λίγο όπως επίσης ε, να ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία των συναδέλφων μου για να εργαστούμε πάνω σε αυτό το κείμενο και θα σας πω ότι όλες αυτές οι παρατηρήσεις ε, των συναδέλφων προσπάθησα να τις συνοψίσω και να τις περιλάβω στο έγγραφό μου αυτό. Θα ήθελα να μιλήσω για ορισμένα σημαντικά σημεία αυτού του εγγράφου είναι σημαντική πλατφόρμα, σημαντική βάση ε, αυτή για την στρατηγική του 2020. Θα πρέπει να δούμε την σημασία αυτών των περιφερειών και οι πόλεις θα πρέπει να έχουν μια σημαντική εντολή, μια σημαντική δυνατότητα για να πετύχουν ε, στη στρατηγική του 2020. Επίσης να πω ότι διάφορες πόλεις χρειάζονται καλύτερη υποδομή, περισσότερη υποδομή. Αυτό είναι σημαντικό και σε πλαίσια ανανέωσης, αλλά επίσης και όσον αφορά την τεχνολογία, να έχουμε με κατάλληλες ενέργειες ε, υποδομές όπως είπαμε χρειάζεται να πετύχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο ζωής της πόλης και υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης. Έτσι και δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι ατενίζοντας προς το μέλλον θα πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής σε αυτές τις πόλεις και χρειάζεται να αντιδράσουμε πάνω σε φαινόμενα όπως περισσότερη εγκληματικότητα και περισσότερη ενεργεία σε αυτές τις πόλεις θα πρέπει να δούμε επίσης και τις εταιρικέ σχέσεις. Οι εταιρικέ σχέσεις αποτελούν σημαντική ιδέα που δεν αναπτύσσεται, δεν αναφέρεται όμως ιδιαίτερα συγκεκριμένα εδώ. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να δημιουργήσει ε, αυτή την υποχρέωση στα κράτη-μέλη ώστε οι εκπρόσωποι από τις αστικές περιοχές να εκπροσωπούνται και επίσης και από τις αγροτικές περιοχές να παρίστανται στην επεξεργασία των ρυθμίσεων στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Και οι δύο λοιπόν θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην οργάνωση, στις δημοσία προγράμματα κλπ. σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνουν, τι συνέπειες όλοι έχουν τα διάφορα μέτρα επιτόπου, αλλά λοιπόν μπορούν να συμμετάσχουν θετικά. Τελευταίο σημείο, σημαντικότατο στην έκθεση αυτή, είναι τα μέσα, τα μηχανικά και αναφέρθαμε το Τζέσικα. Δεν είναι όμως επαρκές αυτό και μόνο. Θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερα χρηματοδοτικά μέσα περισσότερα κονδύλια και, υπάρχει, και θα πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση που να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και ανταγωνιστική απέναντι στα όσα ισχύουν εκεί. Επίσης τα κράτη-μέλη θα ήθελα να τα προσκαλέσω να το ολοκληρώσουν αυτό το Τζέσικα και σε αστικό επίπεδο, εθνικό επίπεδο και περιφερειακό επίπεδο. Θεωρούμε ότι το μέσο αυτό, το εργαλείο αυτό το Τζέσικα θα πρέπει να έχει επιπτώσεις θετικότατες ε, και μακροπρόθεσμα. Υπάρχουν διάφορα θέματα, διάφορες πτυχές όμως που δεν συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση αυτή όπως ε, η τοπική ανάπτυξη, η εκπαίδευση των εκπροσώπων στην ε, δημόσια διοίκηση, στην, αστική, την διοίκηση των πόλεων, επίσης το ούρμπατ, όλα αυτά τι σημαίνουν και ένα πλαίσιο αναφοράς για να είναι μια να υπάρχει μια υφόρο ανάπτυξη σε αυτές τις δομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, δεν υπάρχουν και οι περιορισμοί. Ε, δεν ξέρω ίσως θα μπορούσαμε κάτι να βελτιώσουμε μέσω των τροπολογιών. Επίσης, ανταλλαγή απόψεων έγινε με διάφορους συναδέλφου και συμπεριέλαβα τα διάφορα στοιχεία εδώ. Ερμήνια Μαντσόνη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να επιβεβαιώσω ότι αυτή η εργασία του εισηγητού σίγουρα έλαβε υπόψη τις, τις ιδέες που αναπτύξαμε έστω και πριν από μερικούς μήνες στα πλαίσια μιας συνάντησης με τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δείχνουν ότι έδωσε σημασία ο συντάκτης της έκθεσης αυτής, όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέραμε και το τι έγινε με τα υπόλοιπα που συνέβησαν, όπως είπε και συνάδελφο Βλάσακ, που όλα αυτά που στους Μήνε. Ειδικότερα θα ήθελα να τονίσω μερικά μικροπράγματα, ας τα πω έτσι, και μετά θα υποβάλω και τροπολογίες, κάτι που δεν έκανα μέχρι τώρα, η προθεσμία ισχύει μέχρι αύριο. Εδώ για την εξέλιξη αυτή που, στην οποία αναφέρθηκε ο συνάδελφος Βλάσακ εγώ θα ήθελα από την αρχή στα εισαγωγικά να κάνω μία αναφορά στην πέμπτη έκθεση για τη συνοχή. Εκεί συμπεριλαμβάνεται ιδιαίτερα κεφάλαιο που αναφέρει στο Urban Agenda που δείχνει καλύτερα την γραμμή, των προσανατολισμών που ακολουθούμε στην έκθεση αυτή. Πλήρως συμμερίζομαι το ότι θα πρέπει αυτό το Urban Agent θα πρέπει να ενταχθεί στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής και ότι θα πρέπει να δώσουμε την όθηση, την απαραίτητη στα πλαίσια της στρατηγικής ε, 2020 να τονίσω ακόμα περισσότερο την ανάγκη που υπάρχει να ακολουθήσουμε την πορεία μιας ε, αηφόρων άπτυξης και μιας έξυπνης Ευρώπης ε, ε, τονίζοντας το σημείο 4 τα πράγματα που φαίνεται ότι οι δύο κύριες πτυχές, οι δύο κύριοι στόχοι πάνω στους οποίους επικεντρώνουμε την προσοχή μας αποκλείουν ε, την τρίτη δυνατότητα και θα ήθελα να το δείξουμε αυτό και θα αποτελέσει δε η πρόταση αυτή αντικείμενο τροπολογίες μου εντάξει μπορούμε να υποστηρίξουμε, να τονίσουμε ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη η πολιτική για αστικές περιοχές. Σίγουρα δεν αποκλεί μια πολιτική αγροτικών, των αγροτικών περιοχών και την ανάπτυξή τους ούτε ε, περιφερειακές αστικές περιοχές. Και στο σημείο αυτό καλό θα ήταν να υπάρξει καλύτερη εναρμόνιση ανάμεσα στο σημείο 7 και στο σημείο 10. Εκεί στο πρώτο αναφέρεται οι υποαστικές περιοχές και οι αγροτικές περιοχές αυτές αναφέρονται και μετά και η μεθοδολογία ολοκληρωμένης προσέγγισης αυτής της πολιτικής υπέρ περιοχών που θα πρέπει να εφαρμοστεί κάπως μπερδεμένη με απέναντι σε αυτή την ιδιαίτερη όθηση που δίδει στη γνωμοδότησή του αυτή ο εισηγητής για το μέσο της υποανάθεσης. Την προσέγγιση του εισηγητούν θα ήθελα κάπως να την ε, ε, αλλάξω θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε και ίσως, ίσως να προσπαθήσουμε και σε μερικές περιπτώσεις να έχουμε αυτή την υποανάθεση και να είναι περισσότερο υπεύθυνε τοπικές αρχές σε χαμηλότερο επίπεδο, πιο ειδικό επίπεδο, πιο περιορισμένο και νομίζω ότι με αυτό που φρονώ εγώ αυτό στέκει καλύτερα από τη διατύπωση του εισηγητή. Αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να εκφράσω λίγο πολύ περίπου όλες εκείνες που θα μπορούσαν να γίνουν δεκτές στην οριστική έκδοση της έκθεσης αυτής ε, στα πλαίσια της, ε, των όσων φρονεί και ο κ. Βλάσακ και στα πλαίσια των τροπολογιών που εγώ θα υποβάλω αύριο. Ευχαριστώ, η Κωνσταντσα Κρέλ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Φανταζόμουν ότι υπάρχουν οι οι ηγητέ που να λάβουν το λόγο. Εν πάση περιπτώσει, όμω, θέλω να κάνω κάποιε παρατηρήσει. Θεωρώ ότι είναι και σημαντικό και σωστό. Οπότε μιλάμε για πολιτική, για τις πόλεις να συζητούμε πάντοτε και τη συμπεριλήψη των περιφερειών, της υπαίθρου δηλαδή. Αλλά ταυτόχρονα ε, όταν μιλάμε για πόλεις δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για πόλεις. Άρα Καλά, πολλά και καλά στοιχεία περιέχει αυτή η έκθεση, αλλά συγκεκριμένα προβλήματα, ιδιαίτερα των μεγάλων αστικών κέντρων, Φερρυπίν ότι υπάρχουν συνοικίες χωρίς επαρκείς υποδομές, χωρίς επαρκή ενσωμάτωση στο αστικό κέντρο, ότι υπάρχουν προβλήματα στα μεγάλα αστικά κέντρα τα οποία δεν απαντώνται στα μικρότερα αστικά κέντρα τα οποία δεν τα βλέπει ποτέ η Ήπεθρος, είναι ε, πράγματα τα οποία πρέπει να τα επισημάνουμε, ότι υπάρχουν παραδείγματι πάρα πολύ φτωχές συνοικίες. Και εδώ για να σωματωθεί και μια ευρωπαϊκή πολιτική για τα αστικά κέντρα πρέπει να έχουμε πολύ σαφής, ε, σαφή περιγραφή της κατάστασης Βεβαίω θα πρέπει να επισημανθεί ότι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν την πολιτική τη στρατηγική του 2020 οι πόλει, γιατί μπορούν να επωφεληθούν τα μάλα από αυτήν. επί παραδείγματι το θέμα των μαζικών μεταφορών που θα συμβάλλουν ταυτόχρονα με την ε, επέκτασή τους και στην ε, αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Επί παραδείγματι με την ανάπτυξη μιας διαφορετικής λογικής στην, ε, στο σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική των οικειών στα αστικά κέντρα που επίσης θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής στην, στον περιορισμό της. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία έχει η έκθεση συμπεριλάβει τα δέχομαι, τα υποστηρίζω αλλά θα ήθελα να συμπληρωθούν με κάποιες τροπολογίες. Ευχαριστώ Ρικα Μάνας. Ναι, θα ήθελα ξεκινώντας να συγχαρώ τον εισηγητή για την πολύ καλή εργασία του, πολύ καλή συνεργασία επίσης μαζί του. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι σαν ομάδα και θα το υποστηρίξουμε χωρίς καμία επιφύλαξη. Είναι πολύ σημαντικό για μας και αποτελεί τη βάση εδώ δεν θα πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα και να, να δούμε τι γίνεται σε κάθε λεπτομέρεια αυτό τον αστικό σχεδιασμό. Εδώ επαναλαμβάνουμε όλα αυτά είναι υπέρ της πόλης, το υποστηρίζουμε, δεν μπορούμε τώρα επαναλαμβάνω να μπούμε σε τρομερές λεπτομέρειες. Έχουμε πόλεις στην Ευρώπη που αντιμετωπίζουν εντελώ διαφορετικά προβλήματα και έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πάντω όλα είναι σημαντικά στην πολιτική συνοχή και τη στρατηγική του 2020. Η ε, πολιτική για αστικέ περιοχές ε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε κάθε επίπεδο. Ιδιαίτερα σημαντικό και θετικό είναι ότι όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη θετικά στην έκθεση και επίσης η σχέση, ο σύνδεσμος ανάμεσα στην αστική και στην αγροτική περιοχή. Ε, προς τα εκεί θέλουμε να προχωρήσουμε. Είναι μια πολιτική που υποστηρίζει και τις δύο διαστάσεις και την αστική και την αγροτική. Επίσης σημαντικό είναι να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε μια έξυπνη ανάπτυξη μια υφόρο ανάπτυξη και στις ε, μεταφορές, ε, μια πράσινη πολιτική, να τα υποστηρίξουμε όλα αυτά αποτελεσματικά, ε, τις αστικές περιοχές επαναλαμβάνω στην ανάπτυξή τους και επίσης για την ε, διασταυρούμενη υποστήριξη και αυτή έχει σημασία στον διασταύρωση κονδυλίων. Έτσι θα μπορούσαμε να πετύχουμε καλύτερη χρηματοδότηση και καλύτερη ανάπτυξη σε όλες τις αστικές περιοχές. Πάντως επαναλαμβάνω σε γενικές γραμμές μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το κείμενο αυτό. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και ευχαριστώ τον συγγετή για την συνεργασία. Θα ήθελα να επισημάνω κάποια στοιχεία τα οποία θεωρώ πολύ σημαντικά. Έχουμε καταρχάς κατεπίκουσα ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι ένα πράγμα. Θα πρέπει δηλαδή οι πόλεις, τα αστικά κέντρα, <clears throat> και εσείς αναφέρετε ότι τα αστικά κέντρα παρουσιάζονται ως ε, μοχλή ανάπτυξη. Εγώ όμω θα απαντήσω ότι ο αγώνα για την κλιματική αλλαγή θα διεξαχθεί μέσα στι πόλει, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Επίση, όταν μιλούμε για μοχλού ανάπτυξη, είναι σαν να έχουμε πόλεις δύο ταχυτήτων, αυτέ, οι οποίε είναι ανταγωνιστικέ δηλαδή και είναι μπροστά και εκείνε που, έχουν, που είναι στο πίσω μέρο του σειρμού. Αλλά αυτό είναι σφαλμένο και δεν λαμβάνει υπόψη και τη διάσταση ε, των ε, αστικών κέντρων, τη διαμόρφωση δηλαδή, των αστικών κέντρων που έχουν να κάνουν και με οικονομικούς φυσικά όρους αλλά και με κοινωνικούς και με περιβαλλοντικούς. Είναι λοιπόν σημαντικά τα αστικά κέντρα, αλλά ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχουν πιο πολλέ ανισότητε, φτώχεια, προβλήματα, εκεί που εγκαθίσταται η φτώχεια, με διάφορε μορφέ, με τον αποκλεισμό τον κοινωνικό, με, ε, με τα προβλήματα στροφοδοσία ενεργειακά, με κρίση ω προ τη στέγη, με ανεργία και πολλά άλλα προβλήματα, εκεί είναι οι μεγάλε προκλήσει. Επίσης θεωρώ ότι δεν αρκεί να λέμε βιώσιμη ή αηφόρος πόλη, δεν αρκεί να λέμε πράσινο χρειάζεται παντού. Όχι, συγκεκριμένα. Τι σημαίνει αυτό, δεν υπάρχει μαγική συνταγή για μια βιώσιμη πόλη. Φορετικές η μία πόλη από την άλλη. Τι κριτήρια όμως θα πρέπει να προβάλλουμε έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό τον επιδιωκόμενο στόχο της βιώσιμης της αηφόρου πόλης. Αυτό πρέπει να βγει στο κείμενο. Επίσης, πολιτική συνοχή, ο ρόλο πολιτική συνοχή και ιδιαίτερα υπογραμμίζεται η, ο ρόλος μπορεί να παίξει ως παράγον συνοχής η πόλη, δηλαδή την ε, άρση του αποκλεισμού των ε, περιοχών εκείνων που βρίσκονται στην περιφέρεια και που είναι αποκλεισμένες, άρση των, της αποστέρησης από ε, ποιοτικέ υπηρεσίες σε καλές τιμές, άρση του αποκλεισμού για λόγους περιβαλλοντικούς ή για λόγους ενεργειακούς ή για λόγους απασχόλησης. Οι προκλήσεις μεγάλες του περιβάλλοντος που είναι η ρήπανση, που είναι η συμφόρηση, που είναι η εξάπλωση των αστικών κέντρων είναι ακριβώς η προκληση μεγαλες του περιβαλλοντος που ειναι η ρηπανση που ειναι η συμφορηση που ειναι η εξαπλωση των αστικων κεντρων ειναι ακριβως οι στοχοι που θα πρέπει να προβληθούν. Η πολιτική συνοχή επίσης δεν πρέπει να σχεδιάζεται κατά τρόπον ξεχωριστό. Η αποκλειστικό, αλλά σε συνδυασμό με τις λοιπές πολιτικές, των μεταφορών του περιβάλλοντος, της ενεργειακής, όλα αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν μεταξύ τους για να έχουν μια καλύτερη πολιτική και καλύτερο σχεδιασμό και μεταξύ βεβαίως ε, και στο συσχετισμό μεταξύ της υπαίθρου και των αστικών κέντρων. Ο ρόλος της Ευρώπης θα πρέπει να υπογραμμιστεί φυσικά και ιδιαίτερος οι γενικές επιδοτήσεις για αστικά κέντρα, περιφέρειες που δεν υπογραμμίζονται αρκετά, δεν προβάλλονται αρκετά μέσα από την έκθεση να αποτελούν σημαντική ε, προϋπόθεση για την επιτυχία ενός τέτοιου προγράμματος. Ταυτόχρονα οι σχέσεις οι εταιρικές θα πρέπει να διευρυνθούν για να συμπεριλάβουν όχι μόνο τους παράγοντες πλευράς από φάση τοπικό επίπεδο, αλλά κάθε έναν από τους φορείς που αναπτύσσουν δραστηριότητες στο τοπικό επίπεδο, στην κοινωνία των πολιτών καλύτερα. Θα διατυπώσω λοιπόν πολλές τροπολογίες από ό,τι φαίνεται και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν βλέπουμε το Urban Ferripin. Προγράμματα δηλαδή τα οποία έχουν φέρει καλά αποτελέσματα. Είναι καλή η έκθεση και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε κύριε Τασλάκ να είναι πολύ πολύ καλύτερη. Θα σας βοηθήσω λοιπόν, ελπίζω, με τις τροπολογίες. Ευχαριστώ, Γιάννα Ολμπριχτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η αστική πολιτική είναι μία από τις σπάνιες πολιτικές που διεξάγονται σε τοπικό επίπεδο οι υπόλοιπε πολιτικές επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο τομέα, όπως για παράδειγμα μεταφορές, κλίμα κλπ. Όμως η αστική πολιτική επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο τόπο και επομένως ε, είναι, έχει μια πολύ σημαντική ε, θέση και στο πλαίσιο των συνθήκων. Μιλήσαμε μέχρι τώρα και για μια άλλη τέτοιου είδους ε, πολιτική, η πολιτική των ε, περιοχών της υπέθρου. Αν θέλουμε λοιπόν να μιλήσουμε για την πολιτική ανάπτυξη της υπαίθρου και να τη θεωρούμε πολιτική ε, ευρωπαϊκή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους ίδιους όρους και για την αστική πολιτική. Και γι' αυτό δεν θα συμφωνήσω με τον εισηγητή. Προτείνω λοιπόν να συνεργαστούμε στο πλαίσιο του Urban, γιατί θα μπορούσε το ζήτημα αυτό να επαφίεται μεν ε, στις ε, ε, εθνικές αρμόδιες αρχές, όμως έχει και μια ευρωπαϊκή διάσταση. Αν λοιπόν η αστική πολιτική είναι ένα τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτικής, πρέπει να την αναλάβουμε αυτή την ευθύνη. Διαφορετικά πρέπει να την αφήσουμε εξ ολοκλήρου στις κυβερνήσεις, ε, δηλαδή να λαμβάνει η χώρα η πολιτική αυτή σε εθνικό επίπεδο και μόνο. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε κατά πόσο είναι λοιπόν μια ευρωπαϊκή πολιτική η αστική πολιτική και αν είναι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις ευρωπαϊκές ε, πόλεις δεδομένου ότι προετοιμάζεται το Cities of Tomorrow, πόλεις του αύριο από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε κάτι άλλο ευχαριστώντας τον κύριο Βλάσακ. Παρακαλώ, παρακολουθήστε το θέμα της συγκεκριμένης έκθεσης. Δεν μιλάμε μόνο για την ανάπτυξη των πόλεων μας. Πρέπει να δούμε τη σχέση μεταξύ της αστικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής. Αυτό είναι το θέμα μας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έκθεσης. Δηλαδή, με την έννοια του αστικού πληθυσμού και της αστικής διοίκησης. Πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε τι γίνεται σε ε, επίπεδο πόλεων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αυτή η παρακολούθηση του συγκεκριμένου στόχου. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η σύνδεση που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Ο κύριο Σίμων, έχω καταρχά να ευχαριστώ τον εισηγητή, αλλά έχω και κάποιε παρατηρήσεις, ιδιαίτερη πρωτοβουλία για το mainstreaming του Urban. Νομίζω είναι πολύ σημαντική ω προ την διάθεση των κονδυλίων. Έχει βοηθήσει τη, διάθεση των, τη βελτίωση της αθεσιμότητα των κονδυλίων, αλλά ω προ το περιεχόμενο η εφαρμογή του mainstreaming δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη όπω θα έπρεπε. Έτσι ώστε να βοηθήσει σε μια αηφορία. Και γι' αυτό πιστεύω θα πρέπει να δώσουμε έμφαση ιδιαίτερα για το 2014 και επέκεινα για την υποχρεωτική ενσωμάτωση αυτής της ιδέας. Επίσης, πολύ σωστά επισημαίνεται πως ε, θα πρέπει να ε, συμμετέχουν και οι αιρετοί εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων ε, και των Δήμων στην λήψη των αποφάσεων. Συμφωνώ σε αυτό, λόγω θα πάω ένα βήμα παραπέρα, ότι θα πρέπει δηλαδή να είναι δεσμευτική η παρουσία του ε, στη λήψη των αποφάσεων, στην εξέλιξη των προγραμμάτων, γιατί μερικέ φορέ παραγνωρίζεται η σημασία του. Επίση, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δεσμευθούν για την ανάπτυξη των αστικών κέντρων ως ένα στρατηγικό πρόγραμμα και προκαταβολικά ως προς την επεξεργασία των εθνικών στρατηγικών πλαισίων που θα πρέπει να υποστηριχθούν και πάλι. Και σε ένα πράγμα θα διαφωνήσω μαζί σας, δεν μπορώ να σας ακολουθήσω η ιδέα της πόλης της ίδιας του αστικού κέντρου. Αντιλαμβάνομαι τι διαπροβλήματα βλέπετε, διαπιστώνετε όταν προσπαθεί κανείς ε, να ε, βρει στατιστικά στοιχεία, τα επισημαίνεται άλλωστε μέσα στην έκθεση. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει δυσκολία προς τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τον ορισμό. Αλλά εάν θέλουμε να προσδιορίσουμε, όπως βλέπω ότι προσπαθείτε να κάνετε εσείς το αστικό κέντρο ως αποδέκτη πόρων, οφείλουμε και για το κράτο μέλο, αλλά κυρίω για του φορολογουμένου, να εξηγήσουμε τι ακριβώ εννοούμε με το αστικό κέντρο. Δεν αρκεί λοιπόν να λέμε αστικά κέντρα ή πόλει. Νομίζω ότι μπορούμε να το σκεφτούμε λίγο περισσότερο σε συνεργασία και με τις ενώσεις εκείνες οι οποίες ασχολούνται με τη χωροταξία, ε, ώστε να βρούμε μια προσέγγιση λειτουργική που θα μας απαλλάξει από προβλήματα τύπου πληθυσμός, μέγεθος, έκταση, αλλά θα μας ορίσει ένα λειτουργικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούμε να εντάξουμε την έννοια της πόλης του αστικού κέντρου και που ταυτόχρονα θα μας αφήνει ένα αρκετό περιθώριο ώστε να μπορούμε ε, να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη τα πιο συγκεκριμένα, τις πιο συγκεκριμένες διαστάσεις ή τα υποσύνολα που θέλουν ε, να τα επιλέξουν εκείνα για το, Ευρω... για το αστικό κέντρο. Ευχαριστώ. Κύριος Τσέλερ, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε. Έκθεση πρωτοβουλία αυτή για την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο ευρωπαϊκό αστικό περιβάλλον και το μέλλον στο πλαίσιο τη πολιτική συνοχή. Ε, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει η ανάπτυξη των αστικών κέντρων να συζητηθεί διεξοδικά και εντατικά μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για άλλη μια φορά και ω εκ τούτου Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν αντιλαμβάνομαι τα επιχειρήματα κάποιων συναδέλφων που, ορισ... που σε ορισμένο βαθμό τουλάχιστον ε, με τρόπο ψηφοδεί σχεδόν να αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό του αστικού κέντρου. Δηλαδή φοβούνται να το αγγίξουν. Εδώ και κανένα δύο χρόνια που είμαι εδώ στο Κοινοβούλιο, ένα πράγμα έχω μάθει ότι το αστικό κέντρο και ότι μάλλον η ύπεθρο ε, και το, η ανάπτυξη τη υπαίθρου είναι αυτή που έχουν που έχει το μεγαλύτερο και το ισχυρότερο λόμπι μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό φαίνεται ότι μερικέ φορέ παραγνωρίζουμε και τα αστικά κέντρα. Βλέπουμε ότι 6,1 6,1% της πολιτικής συνοχής μόνο αφιερώνεται στην ανάπτυξη των αστικών κέντρων από τα κονδύλια. Ενώ τα μισό περίπου για την ανάπτυξη υπαίθρου και την αναζωογόνηση της ε, υπαίθρου. Δηλαδή και πάλι μέσα στα αστικά κέντρα το ίμιση e πάει στην ε, ανάπτυξη της υπαίθρου μέσα στα αστικά κέντρα. Η κυρία Κρέλο, ο κύριο Σούλμπριχτ ανέφεραν τα σχετικά με τη στρατηγική του 2020. Θα ήθελα να επισημάνω στου εγώ ότι ό,τι είναι να κάνουμε για τη στρατηγική 2020 θα το κάνουμε μόνο χάρη στα αστικά κέντρα. Είτε πρόκειται για καινοτομία, για έρευνα, είτε πρόκειται για εξασφάλιση ε, ενέργεια ή για αποτελεσματικότητα στην κρίση ενέργεια. Ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε μέσα από τα αστικά κέντρα ή φερειπίν αν θέλουμε να μειώσουμε τον αριθμό των παιδιών που εγκαταλείπουν προώρα το σχολείο. Αυτά θα πρέπει να τα θέσουμε στο επίκεντρο της πολιτικής μας, της περιφερειακής πολιτικής, της πολιτικής συνοχής, δηλαδή το αστικό κέντρο. Διαφορετικό, δε, διαφορετικά δεν πρόκειται να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, είναι σαφές. Γίνεται λόγος επίσης για λειτουργικά προγράμματα, για εθνικά προγράμματα. Εμείς διαπιστώνουμε στη Γερμανία ότι μπορεί να έχουμε πολύ ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση ένα, Τα δε προγράμματα για την περιφερειακή ανάπτυξη βρίσκονται σε επίπεδο διαχείριση στα κρατήδια, στι τοπικέ κυβερνήσει δηλαδή. Πλην όμω τα αστικά κέντρα πάλι είναι στο περιθώριο. Πάλι παραγνωρίζονται, πάλι δεν λαμβάνουν αρκετή προσοχή. Αυτό λοιπόν πρέπει να επιδιώξουμε περισσότερο. και θα προσπαθήσουμε με τις τροπολογίες μας να προσαρμόσουμε την έκθεση. Η Πρόεδρος, ξέρω ότι δεν είναι ευγενικό να στο από το τελευταίο μιλητή να είναι σύντομος, αλλά αναγκαστικά το κάνω. παρακαλώ. Πολύ σύντομα. Φανίστε, Λουρόι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ βρίσκω ότι είναι πολύ εξισορροπημένη η έκθεση του κυρίου Πλάσακ, του συναδέλφου μας. Όμως, πιστεύω πρέπει να είμαστε λίγο πιο φιλόδοξοι σε θέματα πολιτικής ε, συνοχής και αυτό νομίζω ότι θα φανεί και στις διάφορες τροπολογίες. Η αστική ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική βέβαια για την οικονομία, ειδικότερα όταν πρόκειται για νέα ανάπτυξη, για γνώσεις, ε, τεχνολογίες εχμής ε, και για όλα αυτά. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ιδιαίτερα το σημείο 6, δηλαδή το ρόλο των πόλεων στην ανάπτυξη αυτή. Κάποιοι λένε ότι θα έπρεπε να γίνει σε εδαφικό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο, ε, ότι πρέπει να είναι εθελοντικό. Όμως υπάρχουν και ιδιαίτερες περιστάσεις, στις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη. Είναι μοχλή ανάπτυξης η πόλη και συνεπώς κατά την επεξεργασία των προγραμμάτων πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις πόλεις. Όμως νομίζω ότι πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, γιατί έχει γίνει αποκέντρωση σε μερικά κράτη-μέλη, υπάρχουν πόλεις που διαχειρίζονται τα δικά τους προγράμματα και επομένως μπορεί κάλλιστα να γίνει αυτό ε, που θέλουμε να επιτύχουμε σε ένα επίπεδο συνενετικό. Δεν είναι καθόλου αδύνατο κάτι τέτοιο, αντιθέτως αυτό αναφέρει και το σημείο 6. Και ο κύριος Βλάσακ ε, αναφέρεται λίγο στην καθυστέρηση ορισμένων ε, αστικών προγραμμάτων σε, σε εθνικό επίπεδο, όταν βλέπουμε για παράδειγμα κάποιες μητροπόλεις πώς εξελίσσονται. Υπάρχει ο στόχος 3. Μιλάμε για 7% του στόχου 3 και θα ήταν χρήσιμο να λάβουμε υπόψη τις εμπειρίες, τις ανταλλαγές απόψεων και τα κοινά προγράμματα που ε, έχουν λάβει χώρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό τι είναι τελικά μία πόλη. Μήπως πρόκειται για μία Μητρόπολη, μήπως πρόκειται για μία ε, πόλη-περιφέρεια, ε, δηλαδή μία περιφέρεια που ουσιαστικά αποτελεί μία πόλη. Χρειαζόμαστε κάπως έναν πιο συγκεκριμένο ορισμό που θα μας δώσει τη δυνατότητα να διαφωτίσουμε καλύτερα την ε, πραγματικότητα που συνιστά ε, η αστικοποίηση διαφορετικά. Θα το χάσουμε το παιχνίδι και νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να τονίσουμε το θέμα του στόχου 3. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να τονίσω ότι η συζήτησή μας γύρω από τα μελλοντικά ε, αστικά προγράμματα και προγράμματα για την Ήπεθρο, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο συνεκτική. Οι πόλεις συμπεριλαμβάνονται στη διάσταση της ανάπτυξης της υπαίθρου, γιατί η πόλη μπορεί να έχει μία θετική συνέπεια για την ανάπτυξη της ε, Ήπεθρου. Συνεπώς, όταν μιλάμε για πολιτική συνοχή, χρειαζόμαστε κονδύλια στην αστική ανάπτυξη, κυρίω ε, για την ε, άμβλυνση των ε, ανισοτήτων για, τα οποία, για τις οποίες μίλησαν η κυρία Κρέλ και ο κύριος Ολμπρίχτ γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα ε, ποιότητας ε, της ζωής στις πόλεις. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους και πρέπει να πω ότι είναι πολύ σημαντική και η επιρροή της ε, ε, αστικής πολιτικής ε, και, και στην Ήπεθρο. Ακόμα και στα νησιά, στις νησιωτικές περιοχές. Γι' αυτό θα ήθελα να προσανατολίσουμε πολύ περισσότερο τα αναπτυξιακά, τα προγράμματα αστικής ανάπτυξης ή ανάπτυξη της Ήπεθρου στις υπηρεσίες εγκύτητας στις ζώνες υπαίθρου λόγω της εγκύτητας με τις πόλεις ε, μπορούν να παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές. Στην πόλη ε, λαμβάνουν χώρα πολιτιστικά προγράμματα, προγράμματα υποδομών ε, και χάρη στην ύπαρξη της πόλης ε, μπορούν ε, μπορεί η Πεθρός να αναπτυχθεί, οι περιφέρειες να αναπτύξουν ε, τις δικές τους υποδομές. Διαφορετικά, οι δύο πολιτικές οι οποίες είναι τόσο αποκλίνουσες σήμερα, δεν θα βελτιώσουν το βιωτικό μας επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για αυτή τόσο επικοδομητική συζήτηση. Να πω ότι αυτή, σε αυτή την έκθεση βέβαια δεν μπορέσαμε για λόγους χώρου να συμπεριλάβουμε κάθε στοιχείο όπως το είπαμε. Η κυρία Μαντζόνη ζήτησε να συνδυαστούν όλα αυτά με την ε, πέμπτο πρόγραμμα συνοχής. Βέβαια υπάρχει ένας συνδυασμός, ε, θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε τα στοιχεία αυτά. Το ίδιο ακριβώς όπως ε, επιθυμεί και η κυρία Καριντέλη να συνδυαστεί με το Urban και με τα σχετικά προγράμματα. Ναι, θεωρώ ότι υπάρχει αυτός ο συνδυασμός στην έκθεση έστω και αν γιατί θα ήταν λάθος να περιορίσουμε το περιεχόμενο εδώ θα ήθελα να βελτιώσω και εγώ την έκθεση αυτή με όλες τις τροπολογίες που θα έρθουν στα χέρια μου τελικά και θα δούμε και για τις προσεχείς διαπραγματεύσεις τι μπορούμε να κάνουμε για να συμπληρώσουμε να καταλήξω λέγοντας ότι όλοι μας αναρωτιόμαστε τι ακριβώς είναι μια πόλη, ποια προβλήματα απασχολούν μια πόλη. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για πολύ για τα προβλήματα που επηρεάζουν αυτές τις πόλεις. Αλλά στο μέλλον χρειάζεται να εργαστούμε πάνω απ' όλα σε σχέση με το τι είναι οι περιφέρειες γενικά. Δεν μπορούμε να χάσουμε την σχέση αυτή με την περιφέρεια ούτε εδώ σε αυτή την έκθεση γι' αυτό χρειάζεται να στοχεύσουμε σωστά και ε, ο τελευταίος ομιλητής υπενθύμησε πολλά σημαντικά πράγματα πολλές φορές ακριβώς οι πόλεις για την ενέργεια και οι άλλες υπηρεσίες εξαρτώνται από την περιφέρεια και από αγροτικές περιοχές εδώ χρειάζεται λοιπόν αυτός ο συνδυασμός, αυτός ο συσχετισμός και θεωρώ ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για να συμπεριληφθούν αυτά. Αλλά είναι τόσο ευρύ το θέμα. Χρειάζεται βέβαια να είμαστε όλοι ενωμένοι για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, δεν σας είδα και νόμιζα ότι ήθελε η κυρία Κρέλη να πάρει το λόγο εκ μέρου των σοσιαλιστών ως και δυσυχήτρια. Αλλά θέλετε κι εσείς να πάρετε το λόγο, κυρία Κρυσολίνα. Να έχετε το λόγο. Λυπάμαι, λυπάμαι που μπερδευτήκαμε κάπως. Ιδιαίτερα εκτίμησα την έκθεση και Νομίζω ότι έγιναν δεκτές αρκετές προτάσεις και δικές μου αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Θα επιμείνω, θα δούμε με ποιο τρόπο και μέχρι αύριο με τις τροπολογίες πώς να εργαστούμε πάνω σε τέσσερα θέματα στα οποία να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Εδώ αυτή τη συζήτηση που ξεκίνησε για τον ε, ορισμό της αστικής ε, ε, περιοχής. δεν θα ήθελα να σε μια διαπίστωση δυσκολιών επειδή υπάρχουν πάρα πολλές εμπειρίες παρόμοιες στην Ευρώπη. Χρειάζεται να μπορέσουμε να προσφέρουμε και ένα προσανατολισμό σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακόμα κάτι να επιμείνω ότι θα πρέπει οι τοπικές αρχές να συμμετάσχουν περισσότερο και καλύτερα αστική πολιτική δεν μπορεί να προχωρήσει αν ε, δέχονται μόνο προτάσεις και πρωτοβουλίες που έρχονται από αλλού, από ψηλά. Χρειάζεται να μπορέσουν να συμμετάσχουν αμεσότερα ακριβώς οι πρωταγωνιστές ε, της συγκεκριμένη αστικής πολιτικής ε, στο θέμα αυτό, επαναλαμβάνω. Και ακόμα δύο πολύ σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, ο κοινωνικός ρόλος των πόλεων. Και επειδή τώρα τα τελευταία δύο-τρία χρόνια αντιμετωπίζουμε μία κράση και οι ανισότητες αυξήθηκαν, αλλά αυτό ότι υπάρχουν δυσκολίες, ότι είναι φτώχεια, όλα αυτά μας απασχολούν. Θα πρέπει στις πόλεις να το προσέξουμε αναφέροντας το σε αυτή την έκθεση και με πολιτικές που μέσω ενός κατάλληλου σχεδίου, αστικού σχεδιασμού να έχουμε καλύτερες πολιτικές, να δούμε και για διάφορες μειονεκτικές κατηγορίες πολιτών να τους προσέξουμε περισσότερο και ακόμα η διάρκεια που έχει σημασία για την πολιτική του 2020 περισσότερο από μια πολιτική ανάμεσα στην αστική και στην περιφερική πολιτική να θέσω αυτό το θέμα ότι οι ευρωπαϊκές πόλεις χρειάζεται όλο ένα λιγότερο να κανιβαλίζουν ε, αγροτικές περιοχές θα πρέπει να αναγεννηθούν αυτές οι αγροτικές περιοχές και όχι να διαβρωθούν αυτό. Και επίσης βέβαια χρειάζεται να δούμε την ενέργεια, την ανεώσιμη, τις μεταφορές, όλα αυτά. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο γιατί ήδη αρκετοί ομιλητές αναφέρθηκαν σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι η προθεσμία των τροπολογιών ε, είναι 15 Απριλίου 12 το μεσημέρι, 15 Απριλίου 12 το μεσημέρι. Περνάμε τώρα στις εκθέσεις του Ελίωρο και θα ήθελα να του δώσω το λόγο. Δυστυχώς δεν έχουμε όλο το χρόνο που θα θέλαμε, οπότε θα, είμαστε, θα χρειαστεί πάλι να είμαστε σύντομοι. Έχει το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. 4 Δεκεμβρίου μας πέρασε ο κ. Σέματ που ασχολείται με θέματα ακριβώ και φορολογικά μας ενημέρωσε για την υιοθέτηση από τους επιτρόπους της έκθεσης επιτροπής για τα προϊόντα τα οποία δεν τύχουν απαλλαγή σημείωση της φοράς θάλασσης Γουαδελούπη, Γουιάννα, Μαρτινίκ και Ρενιό. Η νέα έκθεση και υιοθέτησή της από την Επιτροπή, αυτό συνέβη μετά από την παρουσίαση από τη Γαλλία μιας έκθεσης ενδιάμεση για αυτά τα προϊόντα και απαλλαγέ και μείωσει. Και επίσης ακολούθησε μια πρόταση απόφασης από το Συμβούλιο που αυτές τις μέρες συζητάμε ακριβώς με 50 ακόμα περισσότερα προϊόντα για την, προϊό, για την Γουιάννα, για αυτά τα προϊόντα που αντιμετωπίζουν διαφορετική φορολόγηση δασμούς ακριβώς βάσει του και του καταλόγου των γαλλικής κυβέρνησης στα βάση του άρθρου 239 άρθρο του συνθήκη που επιτρέπει μετά από πρώτες επίτροπε, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσουμε ειδικά μέτρα για τις υπερπεριφερειακέ περιφέρειες, ακριβώς ε, περιοχές λόγω των ειδικών συνθήκων που επικρατούν εκεί. Αυτό είναι ένα παλιό δασμό που έχει να κάνει και το 1670 ε, από τότε ίσχυσε και από το 1984 και μετά είναι τα περιφερειακά συμβούλια τα οποία παραχωρούν το δικαίωμα αυτό ψηφίζοντα το. Είναι σχετικά με τα πρώτα αυτά, πάει μέχρι και το νόμο του 1992 ε, εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ε, 2 Σεπτεμβρίου του 1989 που έχει να κάνει με τις δασμούς στα τοπικά προϊόντα ώστε όλα αυτά να συνδυασμούν αυτοί οι δασμοί ε, και να συμφωνήσει με την, την μη διακριτική μεταχείριση σύμφωνα με τη ρυθμίση στην Ευρωπαϊκή. Αυτό το 1992 έδειξε ποιοι θα πρέπει να είναι οι όροι για 10 χρόνια για αυτούς τους δασμούς και μετά και πάλι πήγε μέχρι το 1994 από το 1994 για 10 χρόνια που ίσχυσε και η περιφέρεια περιφέρειες έχουν το δικαίωμα να απαλλάσσουν από δασμούς ε, τα τοπικά προϊόντα και αυτό για οικονομική ανάπτυξη τοπική σύμφωνα και αν συμφωνήσει βέβαια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ακριβώς είναι μια μορφή ΦΠΑ. Τα έσοδα δεν πάνε στα κράτη αλλά στις περιφέρειες. Η κράτος εφαρμόζει μειωμένο ΦΠΑ σε αυτέ τις περιφερειακές περιοχές και στις οι περιοχές αυτές συμπληρώνουν αυτό το ΦΠΑ βάσει αυτή τη ρύθμιση τα έσοδα πάνε στι περιφέρειε ακριβώ και είναι 37 και 48% του όλου προπολογισμού των δήμων, των τοπικών αρχών ακριβώ και λοιπά στις περιφερειακέ αυτές Και αυτό ε, τι θέλουμε να κάνουμε αυτό Οπότε η ρύθμιση εξασφαλίζει σε αυτές τις περιοχές έσοδα και τους επιτρέπει οι ίδιες να κάνουν αρκετές επενδύσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξή τους. Και ακόμα αφήνοντα τις διάφορες περιφέρειες να εφαρμόσουν διάφορες απαλλαγές από όπως αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έτσι με αυτές τις ρυθμίσεις ε, προστατεύεται και η ντόπια οικονομία. Είναι πολύ παλιός νόμος, είμαι 1672 σχέδιο και έχει, είναι ζωτική σημασία για την οικονομία, για τι περιφερειακέ κτήσει, αλλά και η διατήρηση του επίπεδου απασχόληση σε περιοχέ ακριβώ που πολλέ φορέ η ανεργία είναι κάπου εκεί κοντά και παραπάνω από το 30%. Γι' αυτού του λόγου θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε του συναδέλφου ότι χρειάζεται ε, τι θα γίνει από το 2013, πώ θα μπορέσουν αυτά τα μέτρα να διατηρηθούν. Και αυτό κάθε 10 χρόνια όλοι οι οικονομικοί παράγοντες εκεί να μπορέσουν να βοηθηθούν γιατί είναι προϊόντα που πάνε στην τοπική αγορά να μην εντοπιτεύσουν ε, να μην ε, υπάρξει μια έλλειψη σιγουριάς, μια βεβαιότητα και οικονομική ουσιαστικά κατάρρευση, καταστροφή οικονομική και κοινωνική. Κύριε Πρόεδρε, αυτά θα ήθελα να πω σχετικά με το θέμα αυτών των προϊόντων και απαλλαγή σημείας φοράς θαλάσσης. Μωρίς Πόγκα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για αυτό το θέμα σχετικά με την εισφορά θαλάσσης. Είναι τεχνική αναθεώρηση των αποφάσεων του Συμβουλίου για το θαλάσσιο δίκαιο ακριβώ και οι υπερπόντιες κτήσεις να προχωρούν σε επιβολή δασμών διαφορετικών από ότι η Γαλλία ή τα υπόλοιπα κάτι μέλη ώστε να ισχυθεί η τα υπολοιπα κρατη μελη ωστε να ενισχυθει η τοπικη βιομηχανια και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά της. Οι αλλαγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβάνουν υπόψη τους καλύτερα τις ανάγκες των περιοχών εκεί που γνωρίζετε όλοι είναι κτίσεις ακριβώς, είναι περιφέρειες ευρωπαϊκές πλήρως για να αντιμετωπίσουμε τον δικό χαρακτήρα της κατάστασής τους μπορούν να υιοθετούνται από το Συμβούλιο ειδικά μέτρα βάσει του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ ακριβώς αυτή η έκθεση το θαλασσιο δίκαιο δείχνει αυτό το ειδικό καθεστώς που εφαρμόζεται σε αυτές τις υπερφερικές ε, περιοχές και βοηθάει αυτές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πατρίς Τυρολιέν. Να ευχαριστήσω ξεκινώντας ε, το συνάδελφο που μας είπε από πώς, πώς και πού ξεκίνησε αυτή η σφορά θάλασσας. Ε, νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στο θέμα αυτό γιατί ο κ. διευκρίνησε ότι αυτό ισχύει μόνο μέχρι το 2014 αν θυμάμαι καλά και μέχρι τότε χρειάζεται να το επανασυζητήσουμε. Αυτό ακριβώς για την εισφορά θάλασσας και το δίκαιο της θάλασσας όπως το είπαμε έχει, είναι ζωτική σημασία για τοπικές παραγωγές ακριβώς και βάσει το άρθρο 349 της συνθήκης αλλά και για τα οικονομικά ακριβώς των τοπικών αρχών που τα έσοδα τους αυτά μπορούν να τα επαναδιανύμουν σε περίπτωση που απαιτούνται κοινωνικές παροχές και μια πολιτική παρόμοια όλα αυτά που σήμερα προτείνονται είναι αποτέλεσμα αποτέλεσμα ιδιαίτερης να ανάμεσα στην Επιτροπή, στη Γαλλία ε, και στην Επιτροπή και δεν πρέπει να καθυστερούμε για την εφαρμογή τους. Γι' αυτό εξ ονόματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών δεν θα προτείνω καμία τροπολογία σε αυτό το σχέδιο ψηφίσματος και σα ευχαριστώ για την προσοχή που μου αφιερώσατε. Ευχαριστώ Ραμόν Μανέσκου από η Κατρίν Γκρέσ μήπω θα ήθελε να λάβει το λόγο τώρα. Όχι, όχι. Κάποιο άλλο κάποιος άλλος που θα επιθυμούσε πάνω στο θέμα αυτό να λάβει το λόγο. Όχι. Τότε μπορούμε να ολοκληρώσουμε την όλη συζήτηση και να σας ενημερώσω ότι ε, ισχύει η προθεσμία τροπολογία πότε είναι 20 Απριλίου στι 12 το μεσημέρι. Σημειώστε το λοιπόν, 20 Απριλίου. Να περάσουμε στην επόμενη έκθεση του Ελιορώ, που είναι για τα ειδικά μέτρα στο τομέα της γεωργίας υπέρ των άκρο απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης. Ελίωρο, έχετε και πάλι το λόγο. Η, τα εδάφη και τα νησιά της Ισπανίας και της Γαλλίας ε, στον ε, Ινδικό ωκεανό ε, είναι οι άκρος απόκεντρες περιοχές, είναι επτά. 30 ε, χρόνια χρειάστηκαν για να ορίσουμε από νομικής ε, απόψεως ε, μια καλύτερη ενσωμάτωση των περιφερειών αυτών στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Πρόκειται για κάτι το οποίο εδρεώθηκε από τη συνθήκη του Άμστερνταμ, άρθρο 279 παράγραφος 2 και η συνθήκη της Λισαμβόνας μέσω του άρθρου 349 επιβεβαίωσε ότι οι άκρος απόκεντες περιοχές σημαίνει μακρύ, μακ, ε, απόσταση από την κοινοτική αγορά και από ειδικέ ε, ε, συνθήκε που φέρνει τι απόκεντε περιοχέ σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο δικαιολογεί την εφαρμογή μέτρων. Ε, το 1989 τα πρώτα ειδικά μέτρα για τις άκρως απόκεντρες περιοχές, περιφέρειες, ε, λήφθησαν από το ΠΟΖΕΗ ένα πρόγραμμα επιχειρησιακό που αφορά ιδιαίτερα τις απομακρυσμένες περιφέρειες και αφορούσε ειδικότερα τον γεωργικό τομέα. Το άρθρο 349 επιβεβαιώνεται έτσι με τα άρθρα 42 και 41 ε, πρώτη παράγραφο, 43 Δεύτερη παράγραφος ε, που θεωρείται η βάση νομική, η νομική, η βάση νομική για την ε, ε ενίσχυση αυτή. Το άρθρο 349 δίνει στην ανάπτυξη της υπαίθρου μία πάρα πολύ σημαντική θέση για την εξέταση κάθε κειμένου που έχει να κάνει με το ζήτημα αυτό. Για ποιο λόγο λοιπόν να υποστηρίξουμε ειδικότερα στις περιοχές αυτές την γεωργία, γιατί ακριβώς ε, είναι ένας οικονομικός τομέας της περιφέρειας αυτές στρατηγικής για δύο λόγους. Ε, πρώτον, ε, γιατί δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και δυνατότητες ανάπτυξης οικονομικής της περιφέρειας αυτές και γιατί η γεωργία και η διαφοροποίηση της είναι τμήμα της ε, επισητιστικής ασφάλειας που είναι πάρα πολύ σημαντική για τις περιφέρειες αυτές, οι οποίες είναι νησιωτικές και μακρινές, απομακρυσμένες από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Οι στόχοι λοιπόν ποιοι είναι. Είναι η αύξηση του βαθμού της ε, ε, ε ασφάλειας που είναι ε, κάτι πολύ σημαντικό για τις περιφερειακές, για τις απόκεντες περιφέρειες και πρέπει ε, αυτή η αυτάρκεια ε, στα τρόφιμα να σημαίνει μείωση των εισαγωγών, ε, μείωση των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων και αύξηση του επίπεδου της ενδογενούς γεωργικής παραγωγής. Για να ε, επιτύχουμε το στόχο αυτό δεν χρειάζεται τις παραδοσιακές παγαλλιέργειες όπως την μπανάνα, τη ζάχαρη και το ρούμι να τις αλλάξουμε με νέες καλλιέργειες. Ε, γιατί όταν οι παραδοσιακές καλλιέργειες πηγαίνουν καλά, τότε ε, η ανάπτυξη γίνεται ακόμη καλύτερη οι παραδοσιακέ καλλιέργειε είναι αυτές που δίνουν τη δυνατότητα της διατήρησης ανταγωνιστικότητας των περιοχών αυτών ε, στην ευρωπαϊκή ε, αγορά ε, και στη... σε σχέση με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και τις χώρες και ε, τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα λοιπόν των παραδοσιακών ε, τομέων ε, πρέπει να μοιράζονται με ισότιμο τρόπο μεταξύ των παραγωγών, των διανομέων και των μεταπίτων για να μπορεί ο καθένας να ζει αξιοπρεπώς βάσει της δραστηριότητάς του από το 1989 όταν άρχισε να ισχύει το πρόγραμμα ΠΟΖΕΙ. Ποιος είναι ο απολογισμός σήμερα. Ο απολογισμός είναι θετικός. Ε, ε, οι έρευνες ε, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2010 απέδειξαν ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή, αυτό το μέσο, όπως επίσης και η ευελιξία του μέσου αυτού, που ε, έχει στεφθεί με επιτυχία. Για μένα είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, ε, επειδή είμαι ο εισηγητή, να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει σε μελέτη αξιολόγηση αντικτύπου κάθε φορά που εμπορικές συμφωνίες ε, διεθνού εμβέλειας υπογράφονται και που οι τομεί τους οποίους υποστηρίζει το ΠΟΖΕΙ μπορεί να απειλούνται. Οι στόχοι λοιπόν του ΠΟΖΕΙ πρέπει να οριστούν καλύτερα και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των άκρος περιφερειακών περιοχών. Και γι' αυτό πρότεινα ένα συγκεκριμένο στόχο που σκοπό έχει την ανάπτυξη της ε, εγχώριας παραγωγής και τη μείωση των εισαγωγών. Επίσης να γίνει διάκριση μεταξύ των ε, προσπαθειών υποστήριξης ε, για, το, για την μπανάνα, το ζαχαροκάλαμο ε, στο πλαίσιο της, των κοινών οργανώσεων αγοράς. Και γι' αυτό ακριβώς να υπάρχει και ένα πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης που μπορεί να ε, υποστηρίξει την ανάδειξη και την ανάπτυξη αηφόρων καλλιεργειών ε, υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ε, κάτι το οποίο πρέπει να αποτελέσει μια νέα διάσταση των στόχων του ΠΟΖΕΙ και το οποίο βέβαια έχει άμεση σχέση με την συνοχή του ΠΟΖΕΗ με την τελευταία ανακοίνωση της Επιτροπής το 2008 όσον αφορά τη νέα στρατηγική για τις άκρος απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης. Ε, για λόγους διαφάνειας, μια, η διαφάνεια που μας απασχολεί όλους, νομίζω ότι είναι σημαντικό οι αιρετοί πρόεδροι των, τοπικών, ε, των αρμόδιων τοπικών αρχών για τα ζητήματα γεωργίας να γνωρίζουν ε, και να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο ε, το ΠΟΖΕΙ, γιατί το τοπικό επίπεδο είναι το επίκεντρο του ΠΟΖΕΙ, οι Ε εκπρόσωποι πρέπει να αναλάβουν ε, το μερίδιο της ευθύνης τους και να γνωρίζουν, να ενημερώνονται από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση ε, με το ΠΟΖΕΙ για τα δύο αυτά επίπεδα. Τα προγράμματα ΠΟΣΕΙ λοιπόν πρέπει να είναι αντικείμενο ε, τακτικής ε, αναθεώρησης βάσει των στόχων που τίθεται στο πλαίσιο του ΠΟΣΕΙ ώστε οι στόχοι που επιδιώκονται να ε, έχουν ως αποτέλεσμα μια πραγματική εφαρμογή των προγραμμάτων. Έχω κάνει πολλές παρατηρήσεις όπως διαπιστώσατε ε, και τροπολογιών και μπορώ, είμαι στη διάθεσή σας βέβαια, να τη συζητήσω με όλους τους συναδέλφους. Ε, δεν είναι γραμμένες στην πέτρα και οι προτάσεις σας ε, θα ε, είναι ευπρόσδεκτες για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε όσο το δυνατόν καλύτερο κείμενο για το ΠΟΖΕ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα σας ακούσουμε τους σκιώδες ηγητές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ξεκινήσω. Πώς. Δίνοντας συγχαρτήρια στον συνάδελφο. Αποτέλεσε άριστη εργασία με ιδιαίτερη προσπάθεια ακριβώς για τη σύνταξη του σημερινού κειμένου που μόλις ακούσαμε, διαβάσαμε. Εδώ να σας πω ότι συμμερίζομαι πολλά από εκείνα που έχει συμπεριλάβει δεν θα ήθελα όμως να είναι μόνο ύμνης αυτών. Εδώ αυτή τη χρονιά συζητήσαμε μια πρόταση για να λύσουμε τεχνικά προβλήματα σχεδόν με χειρουργικό τρόπο απέναντι στον ισχυρό κανονισμό. Και εμείς η Επιτροπή μας η, ε, υπερψήφισε ένα κανονισμό με ε, σχεδόν ε, ομοφωνία, αλλά μετά απέρριψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά είχαν να κάνουν και με το κρασί στη Μαδέρα, με το γάλα στην νησία κλπ. Και μετά λύθηκαν τα προβλήματα. Όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν στην αναθεώρηση του Γενικού κονισμού του ΠΟΣΕΙ. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα που δεν ήρθαν συνολικά σφαιρικά να που τα βλέπουμε ένα-ένα στα πλαίσια του κανονισμού ΠΟΣΕΙ. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν γίνεται να παρακάμψει αυτά τα σημαντικά θέματα και τώρα εμεί δεν μπορούσαμε να βάλαμε τη μητούλα μα εκεί, δεν μας άφηναν. Τώρα όμως είναι η σωστή στιγμή, επανέρχονται πιτάπιτο σε αυτά τα θέματα και αυτά, όπως και τη δεκαετία του 90, για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που απασχολούν ε, μόνιμα αυτές ε, τις υπερ περιφερειακές περιοχές. Ε, οι Κινέζοι <laughs> λένε ότι δεν χρησιμοποιούν κανόνια για να σκοτώσουμε μύγες. Ε, τέλο πάντων, εδώ θα πρέπει να δούμε ίσως υπάρχουν και μύγες που καταστρέφουν τα κανόνια. Θα πρέπει να δούμε αυτές τις μικρές αγορές, τις μικρές ε, άκρος απόκεντρες Είναι το του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Ίσως τα δικά τους τα προβλήματα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τρομερά προβλήματα στην εσωτερική αγορά γιατί θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν παράνομα εμπορεύματα εδώ και εκεί. Ακριβώς επειδή εδώ υπάρχουν λένε ε, για αυτούς τους μικρούς θύλακες θα μπορούσαν ε, να δημιουργηθούν προβλήματα, παρεκκλήσεις, παρανομίες κλπ. Εδώ θα πρέπει να δούμε αυτά τα πράγματα. Βλέπω διάφορες ελλείψεις και στο μέλλον θα προσπαθήσω να διορθώσω τα πράγματα αλλά πώς η Εκτελεστική Επιτροπή επιμένει με τον τρόπο αυτό σε αυτό το θέμα. Εδώ, τα προϊόντα τα οποία μεταποιούνται με πρώτες ύλες που βοηθούνται από το ΠΟΣΕΙ εξάγονται προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε προς τρίτες χώρες βάσει του μέσου όρου 89, 90 και 91. Η Επιτροπή λέει δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τα ποσοστά αυτά γιατί τότε θα μπορούσαμε να έχουμε μια στρέβλωση ε, των εμπορικών ε, κανόνων και οδών. Εδώ με μπερδεύει το πράγμα. Τι γίνεται, είτε τι, τα προϊόντα αυτά θα μπορούσαν να κατακλείσουν την ντόπια αγορά. Κάτι, κάτι δεν καταλαβαίνω, κάτι δεν μου πάει εμένα. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να το λέμε αυτό ότι αυτές οι άκρως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι βιομηχανίες δεν μπορούν να συνεχίσουν την εμπορική τους δραστηριότητα, δεν μπορούν να συνεχίσουν στις εξαγωγές τους γιατί θα πρέπει να περιοριστούν στους μέσους όρους του 89, 90 και 91. Τι γίνεται, θα πρέπει να προσαρμοστεί αυτός ο κανονισμός ε, στις συνθήκες της Λισαβόνας, αλλά να προσαρμοστεί και στη σημερινή πραγματική κατάσταση και εδώ να μπερδεύουμε έτσι αυτές τις μηχανίες. Θα πρέπει να υπάρξει μια εγγύηση μιας κάποιας ευληγησίας και καμψίας για αυτά τα προϊόντα, τα μεταποιημένα με πλήτρες χώρες και όλα αυτά ε, χρειάζεται να υπάρξει ένα πραγματικά ένα πλήρες άνοιγμα θα πρέπει να μετρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά τα τελευταία τρία χρόνια και πέρα από το 1989-1991 να λαμβάνονται υπόψη τα τρία τελευταία χρόνια αν θέλει θα έπρεπε να το συζητήσουμε καλύτερα και με τον εισηγητή. Ήταν κοινή θέση και αντιμετώπιση όλων των βουλευτών από από απόκεντρες περιφέρειες. Εμείς είμαστε λίγοι. Η μόνη λύση μας είναι να παραμείνουμε ενωμένοι και να υπεραμεινθούμε κοινών θέσεων. Αυτό θα κάνουμε και εδώ, αλλά όχι όλα αυτά τα θέματα που έχει να κάνει με αυτές τις δικές μας περιοχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου καταρχάς ε, να συγχαρώ τον συνάδελφο Χουαράου για την εξαίρετη έκθεση. Έχει εντοπίσει τα προβλήματα, τις δυσκολίες έχει προβάλει τις ιδέες του για ένα πρόγραμμα το οποίο γενικά υποστηρίζουμε όλοι. Έχω καταθέσει τις προτάσεις μου για καλύτερη διαβούλευση με τις τοπικές αρχές ως προς τη διαχείριση των προγραμμάτων για καλύτερη αντιστάθμιση δυνάμει της συνθήκης της Γενέβης όπως και ψηφίσει το ψηφισμά του τον Φεβρουάριο φέτος το Κοινοβούλιο στη διαδικασία νομής και της ε, ε, διεξόδους διαφοροποίησης που προτείνονται. Θα ήθελα ωστόσο να επισημάνω θέματα τα οποία μας είχαν απασχολήσει και σε προηγούμενη περίπτωση που συζητήσαμε το κείμενο τη δυνατότητα παραδείγματι για διεύρυνση στη Ρεϊνιόν και τη Μαδέρα της ε, παραγωγής ε, σε άλλες άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες ε, όπως είχαμε προτείνει, θα θέλαμε να σωματιθεί δηλαδή και ξέρω ότι δεν είναι δυνατόν ακόμη αλλά θα θέλαμε με μια καταχώρηση πράξη να, να καταξουδότηση πράξη να έχει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σχετική ρύθμιση να το κρίνει απαραίτητο. Επίση, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πιο ευέλικτη οργάνωση ω προ τι ε, διατάξει που σχετίζονται με την επανεξαγωγή των προϊόντων και τις προμήθειες. Στον εφοδιασμό δηλαδή. Ιδιαίτερα όσον αφορά την αξιοποίηση των κονδυλίων, πρόβλημα βλέπουμε στην προκαταβολική χρηματοδότηση που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο. Ίσως όμως και να ήταν σκόπιμο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να εισαχθεί μια δυνατότητα είτε μέσω συμβάσεως είτε μέσω προεγκρίσεως που θα εγγυάται ε, τη χρηματοδότηση που μπορεί να περάσει μέσα από τραπεζικό σύστημα. Ένα κείμενο λοιπόν που μπορεί να έρθει στο Κοινοβούλιο στα επόμενα πάλι τρία χρόνια θα μπορούσε να έχει νέες προτάσεις, νέες διεξόδους και νέα κονδύλια. Ευχαριστώ κυρία Μάνας. Θα ήθελα να ευχαριστώ εισηγητή για την πολύ καλή αυτή εργασία του και με στοιχεία, πτυχές πολύ θετικές, υποστηρίζει όλα αυτά η ομάδα μου, αλλά ταυτόχρονα θίξω και μερικά προβλήματα που δεν μπορούμε να τα υποστηρίξουμε αυτά. Πρώτα απ' όλα, τι γίνεται. Όπως είπε η συνάδελφος Κρέλ στην ψηφοφορία, θα πρέπει να δούμε τις νέες αρμοδιότητες αυτές, να τις προσέξουμε. Δεν μπορούμε να ε, Φύγουμε όμως και από αυτές. Εδώ έχουμε πράγματα που πάνε πέρα από τις ε, δικές μας ε, ευθύνες. Ε, εδώ σχετικά με την μπανάνα και τη συμφωνία περί μπανάνας. Αυτό δεν είναι στις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας συμφωνία αυτή. Και ακόμα για την εφαρμογή Υπάρχουν θέματα που συζητήσαμε επί μακρόν και επαναλαμβάνω δεν είναι στα δικές μας αρμοδιότητες. Εδώ ε, δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε μια συζήτηση για θέματα που συζητήθηκαν για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, για περισσότερες εξαιρέσεις για αυτές τις, για αυτές τις κτήσεις. Ο συνάδελφος ε, μίλησε για όλα αυτά από κοινού αλλά κάθε κράτος μέλος σίγουρα έχει ένα μέρος του προπολισμού του που διαθέτει σε κάθε παρόμοια κτήση, σε κάθε παρόμοια περιφέρεια. Εάν υπάρξει μια αύξηση από πλευράς Γαλλίας, τότε θα πρέπει να μειωθεί η γραμμή που αφορά τις πληρωμές όσον αφορά τις, ε, ε, τα αγροτικά αλλά είναι θέμα όμως της Επιτροπής Γεωργίας. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν είναι δική μας αρμοδιότητας. Κατά την άποψή μου όμως είναι καλό γενικά το κείμενο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι συνάδελφοι που πήραν το λόγο πριν από λίγο ε, εξέθεσαν πολύ καλά τον δικό χαρακτήρα του προγράμματος αυτού για αυτές τις περιφέρειες και αν ήταν περιοχές εδώ κοντά μας δεν θα το συζητούσαμε γιατί έχουν δυνατότητες παραγωγής οι οποίες εγγυώνται μια ανταγωνιστικότητα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο όμως. Είναι περιφέρειες στη μέση του Ατλαντικού ωκεανού εδώ και εκεί σε διάφορες άλλες υπήρους κοντά. Πολύ μακρινές περιοχές και χρειάζονται ειδικέ σχέσεις λόγω της απόστασης. Αυτό θα μπορούσε να υπερπηδηθεί με πολιτικές που να προσαρμόζουν τα πράγματα σε αυτήν την πραγματικότητα. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε το γεωργικό τομέα. Υπάρχει μια αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ίσες ευκαιρίες που προσφέρονται και εδώ θα πρέπει να εφαρμόζεται. Οι πολίτες των περιφοριών αυτών ε, αντιμετωπίζουν ανισότητες. Παρ' όλα αυτά συμμετέχουν ενεργά στην εσωτερική αγορά. Χρειάζεται λοιπόν μια εγγύηση για όλα αυτά. Γι' αυτό συμφωνώ με τον Σνάφο Τεσέιρα που λέει ότι δεν καταλαβαίνουμε καλά γιατί γίνονται όλα αυτά εδώ οι εισαγωγέ προς άλλες περιοχές πρώτων υλών ε, Εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια εγγύηση για να λάβουμε υπόψη και το κόστος της απόστασης. Μετά όμως ε, δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν εξίσου τον ανταγωνισμό των υπολείπων όταν μεταποιήσουν και πάνε τα προϊόντα σε αυτά και πολύ μακριά και όχι μόνο τοπική τους περιορισμένη αγορά. Παραλαμβάνομαι, αυτό δεν γίνεται αν θέλουμε πραγματικά έναν ανταγωνισμό και αν θέλουμε, όπως ανακοινώνουν εδώ αρκετοί, όπως και ο Επίτροπος Μπαρνιέ, να τους εγγυηθούμε ότι θα συμμετάσχουν πλήρως, όπως λέει και σε ένα εγγραφό του. Εδώ λοιπόν ακόμα κάτι που χρειάζεται το πρόγραμμα αυτό να είναι ευέλικτο, μια κατάλληλη προσαρμογή παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες ε, και κάθε χρόνο χρειάζεται να επεξετάζεται για να δούμε την ευελιξία του αυτή. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν καταλαβαίνω. Πώς δεν μπορεί κανείς να παρέμβει σε μια εμπορική συμφωνία που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα εκεί σε αυτές τις περιοχές. Αυτή η μελέτη επιπτώσεων ακριβώς δεν γίνεται. Χρειάζεται μια παρόμοια μελέτη για να δούμε τι γίνεται μετά από τις αλλαγές της γεωργικής πολιτικής, τι γίνεται σε αυτές τις μακρινές περιοχές να μπορέσει να ενταχθούν κατάλληλα όλα αυτά. Το 2015 τι θα γίνει με τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Θα πρέπει να εξετάσουμε τις επιπτώσεις που θα συμβούν, που θα επηρεάσουν τα πράγματα σε αυτές τις περιοχές. Να ετοιμαστούμε για αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Όλα αυτά αποτελούν δυνατότητα να προσαρμόσουμε αυτά τα προγράμματα και σε εσωτερικής φύσεως γεγονότα αλλά και σε μεγάλα πλατιά παρόμοια εξωτερικά. Έτσι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και μέσω αυτό το προγραμμάτων για να βοηθήσουμε την κατάσταση. Κρέλ. Γκρέσ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Χουαρό για την έκθεση την οποία βρίσκω πολύ εξαντλητική. Φέρει νέα στοιχεία σε σχέση με, την, ε, με τις άκρως περιοχές. Θα ήθελα κάποια σημεία που τα θεωρώ πολύ σημαντικά να υπογραμμίσω. Ε, επί παραδείγματι την έννοια της ασφάλειας σε προμήθεια σε τρόφιμα, δηλαδή αυτάρκεια σε τρόφιμα, στο βαθμό του δυνατού, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, και μείωση των εισαγωγών. Ένα άλλο σημαντικό σημείο στην έκθεση είναι για μένα η προάσπιση των παραδοσιακών πεδίων παραγωγής. Εάν θέλετε, να μην μιλάμε για την παραναπού. που προξενεί αλλεργία στην Φιλανδία. Στην άλλη μιλήσουμε για ρούμι όμως, γιατί μιλήσαμε με τους ε, παραγωγούς ε, πρόσφατα και υπάρχει πρόβλημα και με τον ανταγωνισμό με τη Λατινική Αμερική, Γουατεμάλα, Περού και ιδιαίτερα αθέμει τον ανταγωνισμό των ΗΠΑ που επιδοτούν το, την παραγωγή ρουμιού στις Παρθένους νήσους και το Πουερτορικό. Άρα είναι θέματα αυτά τα οποία πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να μελετήσουμε. Ιδιαίτερα καινοτόμα επίσης βρίσκω την ιδέα οι ε, αιρετοί εκπρόσωποι του λαού να εμπλακούν στις δράσεις που αφορούν το ΠΟΣΕΙ και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να προσθέσω και εγώ δύο στοιχεία που ξέρω ότι δεν είναι καθόλου ε, εύκολο να αντιμετωπιστούν τουλάχιστον το πρώτο από αυτά αλλά πάντως ίσως θα έπρεπε να μιλήσουμε για την ε, γεωργία με παράλληλη ανάπτυξη της διάστασης και των εκπομπών ε, του διοξιδίου του άνθρακα και των κλιματική κλιματικής αλλαγής. Δεν μπορούμε αυτά να μην τα περιλάβουμε. Και επίσης θα σας προτείνω μια τροπολογία για την ενίσχυση της έννοιας της ποιότητας των προϊόντων. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις μου και ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο για τη δουλειά του. Ευχαριστώ θερμά, λέει η Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν θέλετε να λάβετε πάλι το λόγο, κύριε Χώρο. Θα ήθελα ευχαριστώ, να ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο. Ε, οι παρεμβάσεις του ασφαλώς θα μας επιτρέψουν να εμβαθύνουμε στα κείμενα. Ε, συμμερίζομαι τα όσα είπαν οι συναδελφοί τη Τιρολιά και Άλβες για τα προβλήματα σε εξαγωγές των προϊόντων, το πρόβλημα στο γάλα, που μπορεί στη τελευταία ανάλυση να επεκταθεί σε άλλα ε, σε άλλες περιοχές ε, απομακρυσμένες, υπεράκτιες. Επίσης θέλω να την κυρία Κρέας ε, για την ε, συμβολή της στη συζήτηση. Πιστεύω όντως ότι υπάρχει πρόβλημα και στην αναφορά των προϊό, της ποιότητας των προϊόντων αλλά και στο ισοζύγιο διοξιδίου. Για την αρμοδιότητα της Επιτροπής που ανέφερε η συνέλφος Λάνερ, θα ήθελα να πω το εξής, ότι θα πρέπει όντως να επισημάνουμε και να αντιληφθούμε ποια είναι η ουσία του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πρόκειται για ένα άρθρο το οποίο δίνει ένα συγκεκριμένο ρόλο στην Επιτροπή μας, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, ρόλο ηγετικό σε κάθε τομέα, άπαξ και επισημαίνεται ή γίνεται αναφορά στο 349. Δηλαδή πρόκειται για γεωργία, πρόκειται για εμπορικά ζητήματα. Ε, άπαξ και γίνεται επίκληση του 349, πρώτο καθεδρία στην διαδικασία έχει δική μας επιτροπή. Άρα δεν ξεφεύγουμε από το πεδίο αρμοδιοτήτων μας εάν επισημαίνουμε τέτοιου προβλήματα. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. και βεβαίως θα είμαι σε σύνθεση για να μελετήσω όλες τις τροπολογίες που θα κατατεθούν για να καταλήξουμε σε ένα κοινό κείμενο. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Προ... Τροπολογίες 15 Απριλίου, 12 το μεσημέρι. Και επί τη ευκαιρία, παρακαλώ τους αδέλφους από τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, που έχουν άκρως απομακρυσμένες δηλαδή περιοχές, περιφέρειες, να μας επιτρέψουν ε, να μας βοηθήσουν καλύτερα μέχρι το καλοκαίρι, κάπου εκεί στις διακοπές κοντά, να κάνουμε μια μήνυα ακρόαση, γιατί δεν έχουν αντιληφθεί πάντοτε οι συνάδελφοι τι ευθύνε έχουμε για τι άκρω απομακρυσμένε περιοχέ. Όσο γνωρίζετε κι εσεί ότι εδώ υπάρχει μια, ειδική, μια γενική διεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Περιφερειακή Πολιτική που ασχολείται με αυτέ τι ε, περιφέρειε, με αυτήν την ομάδα περιφερειών που έχει δική τη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική και άρα ε, θα πρέπει νομίζω να κατανοήσουμε καλύτερα ποιε είναι οι προκλήσει, ποια είναι τα προβλήματα και οι δυνατότητε και έτσι μαζί με την Γραμματεία και του εν λόγω συναδέλφου θα προσπαθήσω να βρω μια πρόταση για αμήνη ακρόαση. Και δεν θέλω τα τελευταία δέκα λεπτά που έχουμε τώρα να τα αφήσω για τους συντονιστές. Ούτε δέκα δεν έχουν μείνει. Παρακαλώ να αποχωρήσουν όλοι οι λοιποί και να μείνουν μόνο οι συντονιστές στην αίθουσα. Και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα παρακαλώ.